Uh, Ξεκινούμε λοιπόν την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Και πριν περάσουμε στο πρώτο απογευματινό μα θέμα, θα ήθελα να καλωσορίσω εγκάρδια τον Εντάρδο Ραούρ Έλικ, που αντικαθιστά τον κύριο Μπουσόη. Σας καλωσορίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι και ελπίζω να απολαύσετε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 της απογευματινής ημερήσιας διάταξης, την ανάπτυξη του συστήματος e-call σε οχήματα ε, και την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος e-call σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το e-call ε, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ε, προστασίας και ασφάλειας των ε, οδηγών και ε, εντόνως και επιμόνως εδώ και πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε υλοποίηση αυτού του διαλειτουργικού συστήματος και έχουμε επιτέλους κάποια απτή πρόοδο. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγητριά μας, την κυρία Όλγα Σέναλόβα. Καλώς σας απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για το γεγονός ότι επιτέλους μπορούμε να αγγίψουμε στο θέμα του e-call. Και λέω επιτέλους γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένωσε και επιμόνως είχε ζητήσει την υλοποίηση αυτού του συστήματος ε, και εξέφρασε τη λύπη του για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Τελικά τον Ιούλιο του 2010 με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε το ψήφισμα για το e-call με το αριθμό κλίση 112 που θα είναι δωρεάν για όλους τους οδηγούς οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χωρίς άλλους όρους. Και είναι η μόνη λύση για να θέσουμε ένα τέλος στα προβλήματά μας. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση μέχρι το 2015 να εγκαταστήσει υποχρεωτικά το σύστημα e-call μέσω του αριθμού κλίση 112. Και μάλιστα η, η έκθεση με, για την οποία συνεργάστηκα με τον κύριο Κόλλα, τον αρμόδιο εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών, καταλήξαμε σε συμφωνία και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε για πάνω από μία δεκαετία να επιτρέπουμε προαιρετική εφαρμογή του συστήματος, γιατί δεν λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Καταρχήν, το σύστημα e-call δεν μας επιτρέπει μόνο να εντοπίσουμε γρήγορα, αυτόματα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τους κινδύνους, αλλά έχει και άλλα πλονεκτήματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για, τις, για την κατάσταση στους δρόμους, οπότε περιορίζουμε αισθητά τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις και εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Από τον Οκτώβριο λοιπόν του 2015 όλα τα νέα μοντέλα ε, ιδιωτικών ε, αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων θα είναι εξοπλισμένα με το σύστημα e-call και θα δημιουργηθεί και η υποδομή για την σωστή διαχείριση και διαβίβαση των κλήσεων e-call, ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του συστήματος πανευρωπαϊκά. Χαίρομαι γιατί οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα μακροχρόνια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τη θέση σε λειτουργία αυτού του συστήματος που θα έχει σημαντικά ωφέλη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και γι' αυτό θα πρέπει να περιοριστούμε στους ελάχιστους κοινοτικού καλώνες που θα εξασφαλίσουν την λειτουργικότητα αυτού του συστήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε απόπειρα ε, καθυστέρησης της διαδικασίας ε, είναι ανεπίτρεπτη και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας θα δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στη διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πια στη διάθεσή του όλες τις νομοθετικές προτάσεις ε, για το e-call επιτάπητος. Οπότε είναι μοναδική ευκαιρία για να στηρίξουμε αμέριστα αυτό το πολύ χρήσιμο σύστημα και ελπίζω να το πράξουμε. Η δεμή, η ιδέα ενός ασφαλούς συστήματος που θα σώζει 2.500 ανθρώπινες ζωές το χρόνο, ε, θα αναβαγίσει. Θα ακούσουμε σίγουρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρουσίαση, αλλά θα πρέπει να μας ε, ενημερώσει για το πώς θα γίνουν τεχνικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι αυτών των συστημάτων, γιατί δεν είδα κάτι τέτοιο στην πρόταση. Επίσης προσοχή, ε, έχουμε και τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Χαίρομαι πάντως γιατί ήταν αγαστή συνεργασία με τους και και με τον συνάδελφο Ντεμπάκερ. Έχουμε ήδη προλιάνει το έδαφος και νομίζω ότι είναι προς ε, το κοινό μας συμφέρον να διεκπαιρεώσουμε τις εκθέσεις το συντομότερο δυνατόν, ώστε να τις παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια ήδη από το Φεβρουάριο του 2014 και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. πολύ. Ας ακούσουμε λοιπόν σκιώδεις και τους ε, υπευθύνους εκ των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Χάντζελη και έχει το λόγο. Α, συγγνώμη. Δεν είμαι σκιώδης ηγήτρια για το θέμα αυτό. Απλώς ζήτησα το λόγο αργότερα για τη συζήτηση. Συγγνώμη που σας μπέρδεψα. Do we have anyone from the EPP? Από το ΕΛΚ έχετε κανέναν ε, ως σκιώδη γιατί δεν έχω κατάλογο εδώ στις ε, σημειώσεις του Προέδρου. Δεν... <laughs> Και πάλι συγγνώμη. Τελικά ε, εγώ αναπληρώνω τον κύριο Βαντεγκάμπ τον σκιώδη μας ηγητή, οπότε επιτρέψτε μου να μιλήσω τώρα. Συγγνώμη, μου λίγο αφηρημένη και το ξέχασα. Οπότε, όντω, εγώ κανονικά θα έπρεπε να έχω το λόγο, γιατί αναπληρώνω τον εισηγητή μα. Α, δεν είστε οι πρώτοι, συνέχεια μα συμβαίνει, δεν ξέρουμε ποιον αναπληρώνουμε, πού βρισκόμαστε. Α, σα ζητώ και πάλι συγγνώμη. Λοιπόν, θα ήθελα, αξιότιμοι συνάδελφοι, να σα ε, μεταφέρω τη γνώμη του σκιώδου συγγητού του κυρίου Βιμ με παρακάλεσε να διαβιβάσω εδώ τη θέση του. Κατά τη γνώμη του, η υποχρεωτική εγκατάσταση της τεχνολογίας e-call που θα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων ή στη μείωση των μοιραίων ατυχημάτων και στον περιορισμό ή το μετριασμό των τραυματισμών είναι ένα πολύ καλό βήμα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί η ασφάλεια είναι το ζητούμενο και η ύψητη προτεραιότητα και με το e-call θα έχουμε την ευκαιρία να την εξασφαλίσουμε. Ο κύριος Βαντενκάμπ εύσε την προσοχή μας σε μια σημαντική πρόκληση, γιατί ένα υποχρεωτικό σύστημα e-call μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η οδική βοήθεια, η διάγνωση ή κάποιες δραστηριότητες που αφορούν την διατήρηση και την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Συμφωνώ με τον ασκιώδη συγητή μας και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα πρέπει να στηρίζεται σε μια πλατφόρμα που θα είναι ε, προσιτή, δωρεάν και θα λειτουργεί σωστά και με βάση τις αρχές του ανταγωνισμού και την αρχή της ελεύθερης επιλογής των ε, καταναλωτών αλλά και της ανεξαρτησίας των παρόχων υπηρεσιών. Δεν μπορεί ένα σύστημα να μας ε, επιβάλλει που θα πρέπει ο οδηγός να κάνει το σέρβι στο αυτοκίνητο του. Γιατί κάτι τέτοιο θα απέβαινε ει βάρος του ανταγωνισμού. Θα πρέπει πάντως η υποχρεωτική εγκατάσταση του e-call να εξασφαλίσει την προσφορά και εναλλακτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν οι ε, οδηγοί να διαλέξουν τον πάροχο υπηρεσίας τους και με βάση τα στήματα τηλεματικής θα πρέπει να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει αυτούς τους στόχους, γιατί με την ε, μορφή που έχει τώρα δεν εξασφαλίζονται τόσο θεμελιώδη ζητήματα και για τους καταναλωτές, αλλά και για τους ε, εκπροσώπους ε, της ανεξάρτητης αγοράς. Θα πρέπει με τις διατάξεις αυτές να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη επιλογή και την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ένα άλλο θέμα που μας επισημαίνει ο σκιώδης ηγετής ο κύριος Βαντενκάπ και για το οποίο έχει κάποιες ελαφρές επιφυλάξεις αφορά το χρόνο θέση σε ισχύ. Γιατί κατά τη γνώμη, κατά τη γνώμη του κύριου Βαντεγκάπ θα πρέπει το σύστημα αυτό να εφαρμοστεί, να εγκατασταθεί και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι όντω ρεαλιστικό να εγκατασταθεί το σύστημα μέχρι το 2015. Γιατί στην Πολωνία θα έχουμε πρόβλημα. Καλύτερα να περιμένουμε λίγο, αλλά να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά και σωστά, για να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Θα ήταν κρίμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση των δυνατοτήτων κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα μέχρι το 2015. Επίσης, ε, ο κύριος Βαντενκάπ επισημαίνει ότι μερικοί παραγωγοί ήδη έχουν κάποια προηγμένα συστήματα e-call που εξασφαλίζουν επιπλέον πληροφορίες που είναι πολύ χρήσιμες για τα σωστικά συνεργεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ο αριθμός των ροσάκων που χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό το σύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, και προς όφελος των καταναλωτών. Ευχαριστώ και Ζητώ ακόμη μια φορά συγγνώμη για, για το μικρό μπέρδεμα, αλλά θα ήθελα να σας παρουσιάσω, όπως και έκανα, τη γνώμη του σκιώδου συγγητού του ΑΕΚ. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ θερμά. Από τους φιλελευθέρους ποιος έχει αναλάβει ο Σκιώδης. Δεν έχουμε κανένα παρόντα για σχόλιο. Η πράσινη. Η κυρία Ρίολε. Δεν ε, έχω κάτι συγκεκριμένο ακόμη. Θα είμαι εγώ μάλλον σκιώδη συγγήτρια. Θα ήθελα απλώ ε, για την συγγητρία να πω ότι ήμασταν επιφυλεκτικοί ως προς τη δυνατότητα ε, και την ταχύτητα με την οποία θα μπορούσε να εισαχθεί το θέμα. Καλό είναι να υπάρχει πίεση χρόνου, αλλά παρόλα αυτά πρέπει και να αναλογιζόμαστε σε τι αποδιόμαστε και πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ε, το στόχο, πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο της ε, διαλειτουργικότητας σε διάφορες πλατφόρμες. Υπάρχουν διάφοροι φορείς πάροχοι υπηρεσιών όπως λέγονται, οι οποίοι προσφέρουν συγκεκριμένε υπηρεσίες. Θα πρέπει το θέμα αυτό να το συστήσουμε με την Επιτροπή, η οποία μας λέει ότι είναι η, η πρόταση αυτή ε, ουδέτερη. Ε, αυτό πρέπει να επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε σε ποιο βαθμό μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα ε, διάφορα συστήματα. Ε, βάσει της προτάσεώς της. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, αν είναι το χρονοδιάγραμμα ρεαλιστικό. Άλλη μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν επίσης έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια μηνύματα λάβει ενδεχομένω από το Συμβούλιο για το πώς βλέπει το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Φυσικά θα έχει την ευκαιρία η Επιτροπή να αντιδράσει όταν ακούσουμε τους σκιώδεις πρώτα. Συντηρητικοί μεταρρυθμίστες, ο κύριος Χάρμπορ δεν είναι παρόν. Έτερος, που ενδεχομένω μπορεί να... Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα και από την Επιτροπή Μεταφορών, όπου είμαι σκιώδης ηγετής εκ μέρους του ΕΛΚ της πολιτικής μου ομάδας ε, για το θέμα αυτό. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη στενή συνεργασία. Θέλουμε για όλη την Ευρώπη και για όλους τους πάντες την δωρεά, την δωρεάν ανάπτυξη του συστήματος Η Ιδιαίτερη σημασία έχει να μεταβιβάζονται με το σύστημα αυτό ε, στοιχεία καταρχάς για την ομάδα αίματος αλλά και για ενδεχόμενα προβλήματα δυσανεξίας ή αλλεργίας σε φάρμακα ε, εφόσον φυσικά το δέχεται ο ίδιος ο οδηγός. Φαίνεται πολύ φιλόδοξος ο στόχος. Ωστόσο, όσο φιλόδοξος και αν φαίνεται, ίσω περιβαλλοντικά φιλόδοξο δηλαδή, εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο να δράσουμε και να δράσουμε τώρα και να επιδιώξουμε όσο μπορούμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Αν χρειαστεί θα επανέλθω στον κατάλογο των σκιωδών. Από την ΚΟΕ πάλι δεν βλέπω κανέναν. Ούτε από τους ε, από την Ευρώπη των, των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Έτερος. Τότε μπορούμε να κλείσουμε αυτό το μέρος της συζήτησης για να δώσουμε το λόγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Επιτέλους βρισκόμαστε σε μια θέση να συζητήσουμε αυτή την πρόταση για το e-call. Θυμάστε ότι είναι προϊόν του δικού σας οίκου. Όχι μόνο μας έχετε απειλήσει να κάνουμε μια πρόταση, αλλά και στην ίδια την έκθεση πριν από ένα χρόνο, την οποία δείτε πριν από ένα χρόνο, πολύ ρητός αναφέρατε την ανάγκη ύπαρξη ενός εργαλείου απλού, που θα βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνολογία, εύρωστο εργαλείο, χαμηλού κόστους, ε, κάτι περίπου να κοστίζει γύρω στα 40 ευρώ ανά όχημα. Μας ζητήσατε κάτι δημόσιο, μια δημόσια υπηρεσία και μας είχατε πει ότι μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο κάθε οδηγός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα είτε ε, χειροκίνητα να στείλει μια κάνει μια κλίση σε, επίπτωση, σε περίπτωση έκδοτης ανάγκης, είτε αυτομάτως να γίνεται μια τέτοια κλίση. Εφόσον βασίζεται σε κάτι το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά και λειτουργεί πολύ καλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του αριθμού 112. Δεν φεύγουμε λοιπόν από αυτή την αρχή. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αναδείξατε στην έκθεσή σας και βεβαίως ο κύριος Κόχ ε, ε, πρόθεσε αυτή την ιδέα ήταν η ιδέα της ουδετερότητας. Και παρακαλούμε να μην ε, επικεντρωθούμε σε μια τεχνολογία που δεν μπορεί να ε, αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και να μην ε, αποκόψουμε πρωτοβουλία για άλλε υπηρεσίε με προστιθέμενη αξία. Και από αυτή την έννοια η πρόταση που έχετε ενώπιόν σας είναι διαφορετική από αυτή που συζητήσαμε πριν από 7-8 χρόνια, καθώς ε, το τσιπάκι αυτό, αυτή η κάρτα SIM που θα ενσωματώνεται σε κάθε όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το e-call, αλλά σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο ιδιοκτήτης του οχήματο το αποφασίσει, θα μπορούσε να έχει και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Μια ακόμα αρχή είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την ανοιχτή μας προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να, να πούμε λοιπόν ότι δίνουμε την επιλογή στον οδηγό. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει την αυτόματη κλίση 112, ή αν θα έχει μια συνδρομή σε μια πιο εξελιγμένη υπηρεσία υποβοήθησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Να είναι λοιπόν δική του επιλογή. Τουλάχιστον όμως να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε αυτοκίνητο από τον Οκτώβριο 2015 και μετά θα έχει αυτό το μηχανισμό. Σημαντική είναι και μια άλλη πτυχή που έχει υπογραμμίσει η Επιτροπή σας το 70% των οχημάτων σήμερα είναι ε, μεταχειρισμένα. Και χάρη στις δικές σας προσπάθειες, τα περισσότερα από αυτά, όλα είναι και περισσότερα, απολούνται διασυνοριακά. Και έτσι είναι σημαντικό να έχουμε μια εγγύηση που ε, να μας διαβεβαιώνει ότι έχουμε κάτι στο όχημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς υπάρχει ε, και για τους επόμενους μελλοντικού ε, ιδιοκτήτες. Σε ό,τι φορά το χρονοδιάγραμμα, Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό. Έχουμε δύο σκέλη της πρότασης. Την πλευρά των αυτοκινήτων, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα για τους κατασκευαστές να έχουν το προϊόν τον Οκτώβριο του 2015. Υπερθυμίζω ότι δεν θα ισχύει για κάθε νέο όχημα, για κάθε νέο μοντέλο θα ισχύει. Έτσι υπάρχει ένα περιθώριο. Και αν δείτε όλες αυτές τις απίστευτες καινοτομίες που μας ε, προτείνουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στα υφιστάμενα μοντέλα, αυτή η νέα τεχνολογία δεν ε, θα προκαλέσει προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, δηλαδή για τις, οι εθνικές αρχές που θα λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις, όλες οι ενδείξεις είναι θετικές. Έχουμε ακόμα και κράτη-μέλη όπως η Ρουμανία, η Τσεχία, που ήδη είναι πλήρως εξοπλισμένες. Πλήρως εξοπλισμένα τα κράτη-μέλη. Αλλά όλα τα κράτη-μέλη μας αδιαβεβαιώνουν ότι πράγματι εξοπλίζονται. Ουσιαστικά πρόκειται για επικαιροποίηση του λογισμικού που χρησιμοποιούν στο κέντρο έκτακτης ανάγκης και κάποια οργανωτικά ζητήματα και επιλογές για το φιλτράρισμα των κλήσεων. Τώρα για το Συμβούλιο μια φορά το έχουμε πιάσει στον ύπνο το Συμβούλιο. Είναι λοιπόν θετικό. Μια φορά να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να δώσουμε μια θετική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλες απορίες ή σχόλια για το θέμα αυτό. Αλλιώ να επανέλθουμε στην εισηγητριά μας, την κυρία Σενάλογα. Α, βιάστηκα αλλού κοιτούσα. Κυρία Στάινερ. Μετά το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το 2025 ε, για τη θέση ισχύ. Πολύ ε, ενδιαφέρον, αλλά πώς θα εξηγήσετε στον κόσμο ότι και πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα μέσω, ανακράτος μέλος μέσω της αυτοκινητοβιομηχανίας, πώς θα το κοινοποιήσετε, γιατί Ελάχιστοι γνωρίζουν την πρόταση αυτή, που είναι πολύ καλή πρωτοβουλία και ίσως θα πρέπει να την προβάλλουμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να δώσετε απάντηση θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ενθάρρυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει ο ίδιο, οι ίδιοι κατασκευαστές το ταχύτερο δυνατόν να ενημερώσουν την πελατεία τους και να την εξηγήσουν ως ένα πάρα πολύ πολύτιμο πλεονέκτημα πιο, για ένα πιο υπεύθυνο και ασφαλές προϊόν. Και φυσικά θα συνεχίσουμε εμείς κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας για να εξηγήσουμε καλύτερα τι συνεπάγεται. Άρα θα θέλαμε πριν δώσουμε υπερβολικά πολλές διαβεβαιώσεις να έχουμε τουλάχιστον πλευρά του κάποια διαβεβαίωση για το αν μπορούμε να θυρίσουμε το χρονοδιάγραμμα και αν ή ε, ε, μη τι άλλο στις αδρές της γραμμές αυτή η ιδέα είναι αποδεκτή. Αυτό θα θέλω να μιλήσω. Ευχαριστώ όλοι κύριε Πιετικά. Είναι αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Θα παρακαλώ την συγκεκριμένη να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. několik dat. To... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και να σας αναφέρω και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Ιδιαίτερα ως προς τη βιωσιμότητα της πρότασης και το εφικτό του χρονοδιαγράμματος. Το e-call το αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2005. Και έχει περάσει πολύ καιρό έκτοτε και νομίζω ότι έχει οριμάσει η κατάσταση και μπορεί πια η αυτοκινητοβιομηχανία να προβλέψει την ακολουθητέα κατεύθυνση. Έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα για την εξακρίβωση της ετοιμότητας των κρατών μελών και του βαθμού προετοιμασίας τους για την εγκατάσταση του συστήματος e-call στον αριθμό κλίση 112. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πόσο έτοιμα είναι τα κράτη-μέλη και το δυνατότητα προσφοράς ε, από τρίτες χώρες ε, του e-call. Το e-call έχει σχεδιαστεί ως κοινοφελής υπηρεσία αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλες υπηρεσίες που έχουν προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ πάντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τους και ηγητές μας. Και επίσης ευελπιστώ ότι θα φέρουμε σε πέρα στο θέμα αυτό πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Και επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να συμφωνήσουμε το συντομότερο δυνατό και να καταλήξουμε στην εγκατάσταση του συστήματος. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα. Και έτσι θα επανέλθουμε. Σε μεταγενέστερο στάδιο παρακαλώ πάντως ε, και την Επιτροπή μας ε, να συζητήσει σύντομα το θέμα. Κλείνοντας λοιπόν τις συζητήσεις και τα σημεία 10 και 11 στην ημερήσια ταξί μας, παρακαλώ τις πολιτικές ομάδες να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής που έχουν ως εκπροσώπους εδώ, γιατί φαίνεται σήμερα να προχωράμε πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμά μας και καλό θα ήταν να είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους ε, παρόντες, τους ε, υπευθύνου, να τους είχαμε παρόντες εδώ νωρίτερα. Και πάω στο επόμενο θέμα της ημέρας της διάταξης. Έκθεση για μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παύλο Αριάς Ετσεβερία. από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά μια και έχει προβλεφθεί η συζήτηση να ξεκινήσει στις 4, ο κύριος Ατσιβερία δεν είναι εδώ. Διακόπτουμε λοιπόν για 10 λεπτά. Τον έχουμε ήδη ειδοποιήσει, θα χρειαστεί όμως κάποιο χρόνο μέχρι να διανύσει την απόσταση μέχρι την Επιτροπή μας. Παρακαλώ λοιπόν σε 10 λεπτά να είμαστε όλοι πίσω. Ευχαριστώ. <coughs> Να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τώρα. Αφού έχουμε όλους τους αρμοδίους εδώ. Και ας περάσουμε στην ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καθώς αναμένεται να αναπτυχθεί αυτή η αγορά, Ελπίζουμε να αναπτυχθεί αντίστοιχα και η αγορά παράδοσης δεμάτων. Ήρθε λοιπόν ο συνάδελφος, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή. Και είναι πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας καλωσορίσω μετά το καλοκαίρι. Ελπίζω να γυρίσετε ακμαίοι με φορτισμένες μπαταρίες, γιατί το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας θα είναι αρκετά έντονο και γεμάτο. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί το πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων ως προς το σχέδιο έκθεσής μου. Θα ήθελα να εξηγήσω τις αδρές γραμμές της έκθεσης. Η έκθεση αυτή ακολουθεί την κατεύθυνση που είχα ανακοινώσει και τον Ιούνιο όταν έκανα την πρώτη παρουσίαση. Χώρισα την έκθεση σε πέντε τμήματα, οι βασικούς άξονες. Το πρώτο τμήμα αφορά την ανάγκη να έχουμε ποιοτικέ υπηρεσίε παράδοσης, που είναι σημαντικός πυλώνας για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε τον Ιούνιο, διαπιστώσαμε ότι η αγορά και διανομή των ε, αγαθών που αγοράζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι βασικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς και θέλουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ε, προσιτές ε, που θα είναι σημαντικό να στο τμήμα για να προωθήσουμε τις διαδικτυακές αγορές και να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή αγορά. Δεύτερο βασικό άξονα ε, πέραν της, ε, των ολοκληρωμένων υπηρεσιών είναι η ανάγκη να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε ότι η αγορά προσφέρει μια τεράστια γκάμα επιλογών στους καταναλωτές και θα πρέπει να έχουν ελευθερία να διαλέξουν το κατάλληλο. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη τους, να ενημερώνουμε σωστά τους καταναλωτές και να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή από πού αποστέλλεται το δέμα τους, πότε θα φτάσει, ποιος το έστειλε, ποιος είναι ο αποστολέας, ποια θα είναι η τελική τιμή και φυσικά τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επιστροφής και σε ποιο θα πρέπει να απευθύνουν τα παράπονά τους. Τρίτος άξονας επικεντρώνει την προσοχή μας στις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει ε, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες παράδοσης ε, να, να αποτελέσουν εργαλείο και για τις μικροπεσίες επιχειρήσεις για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε ελεύθερο και αποτελεσματικό ανταγωνισμό για να αυξηθεί η προσφορά των υπηρεσιών των παρόχων και να μειωθεί και η τιμή του τελικού προϊόντος. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τεθεί ένα τέρμα στο κατακαιρματισμό της αγοράς και να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, απλές, ε, φθηνές ε, και ασφαλείς υπηρεσίες παράδοσης. Γιατί οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θα πρέπει να χάνουν ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ε, μεγάλες ε, εταιρείε που χρησιμοποιούν καλύτερα το ίντερνετ ε, και δεν θα πρέπει να τεθούν σε δυσμενή θέση. Τέταρτος άξονας, καινοτομία και διαλειτουργικότητα. Νευραλγικοί ναι, παράγοντε, ώστε οι αγορέ παράδοση να προσαρμοστούν στι ανάγκε τη ψηφιακή αγορά. Δεν χρειάζεται να εγκρίνουμε κάποιε ρηξικέ έλευθες νομοθετικέ αλλαγές, γιατί μετά τι ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ζήτηση ούτε από του καταναλωτέ ούτε από τι επιχειρήσει για τη δημιουργία νέων κανονιστικών διατάξεων στον τομέα αυτό. Ήδη έχουμε επαρκή νομοθεσία που απλώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά και πιστά πριν ε, προτείνουμε νέε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Αυτό που οφείλουμε ως ε, νομοθέτες είναι να θαρρύνουμε τον κλάδο να υλοποιήσει τους ε, μέχρι τώρα στόχους χάρη σε συμφωνίες και κοινέ προσπάθειες για προτυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών ε, ή της ετικετοθεσίας για παράδειγμα, ώστε να επωφεληθούμε όλοι από τις αλλαγές αυτές. Η έκθεση προτείνει πολλά μέτρα που βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να προωθήσουμε μία, ένα συμβόλαιο μεταξύ των χρηστών, των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών, ώστε να υλοποιήσουμε τους επιθυμητούς στόχους σε συγκεκριμένο και έφτατο χρόνο. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε, αλλά απλώς να προτείνουμε. Ο κλάδος ε, είναι ικανός ε, να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα, γιατί ήδη υπάρχουν πολλοί άριθμες πρωτοβουλίες για τα συστήματα εύκολης επιστροφής, εντοπισμού και παρακολούθηση της παραγγελίας, καθώς και διαθεσιμότητα θηρίδων παραλαβής των δεμάτων. Και εμείς ως νομοθέτες σε αυτή τη φάση θα πρέπει να παροτρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να καταλήξουν σε συμφωνίες για να επιλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και να ενθαρρύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών παράδοσης να επιταχύνουν τη διαδικασία ανέβρεσης αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ τριών φορέων, των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών επιμελητίας και παράδοσης. Και αυτός ο διάλογος θα πρέπει να επιβλέπεται από τα θεσμικά όργανα, ώστε να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των στόχων μας. Και έρχομαι στο πέμπτο και τελευταίο άξονα της έκθεσης που μιλάει για την ανάγκη της εποπτικής λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων. Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και για το, τη διόρθωση του κατακαιρματισμού, αλλά για την εξασφάλιση του θεμητού ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Αυτή είναι η πρωταρχική άξονες της έκθεσής μου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι σήμερα προτεραιότητά μας είναι να ακούσουμε τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών των πολιτικών ομάδων και γι' αυτό περιμένω με αδημονία τα σχόλιά τους. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πολύ επικοδομητική πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές και εκεί έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για επιμέρους στοιχεία της έκθεσης και θα ήθελα ευκαιρία να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για το συνεργάσιμο πνεύμα τους και την προθυμία τους να βρούμε κοινέ λύσεις προκειμένου να προωθήσουν αυτή τη σημαντική έκθεση στα πλαίσια των πρωτοβουλειών που στόχο έχουν την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις. Σε ένα λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την έκθεσή του, για το σχέδιο έκθεσής του που είναι πολύ αξιόλογο και να τον ευχαριστήσω για τις πρώτες ε, συναντήσεις που είχαμε και για τις επικείμενες που θα έχουμε με τον εισηγητή. Διαπιστώνω ότι ε, με την έκθεση σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες παράδοσης, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η έκθεση επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν και επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών παράδοσης, ε, ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης, της διαφάνειας και ε, αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών τιμών Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και θα πρέπει η πρόσβαση στις υπηρεσίες παράδοσης να επεκτείνεται σε όλες τις ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στις πιο απόμακρες περιοχές. Θα ήθελα να ενισχύσουμε το, τη διατύπωση του σημείου 16 που μιλά για ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Πιστεύω επίσης ότι μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης ε, των θεμάτων. Αυτό το αντικείμενο έχουν και οι τροπολογίες μου. Αν και καταρχήν ε, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τον εισηγητή. Ένα άλλο το θέμα, για να μην πω το ζήτημα για τους σοσιαλιστές, είναι το θέμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των θεμάτων στα πλαίσια βελτίωσης ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν αναλύσαμε λεπτομεριακά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι ως αρμόδια Επιτροπή εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών παράδοσης και των συστημένων δεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναφέρθηκε σε μια ξηρά αρχών, όπως είναι ένα χαρακτηριστικό σήμα ή διακριτικό που θα φέρουν τα δέματα και που θα είναι ένα είδος εγγύησης για τους καταναλωτές η ύπαρξη αυτού του, του σήματος. Και επίσης ε, θα ενισχύεται η ενημέρωση των καταναλωτών και άρα και η αξιοπιστία του συστήματος. Καλό είναι οι υπάρχει τέτοιων υπηρεσιών παράδοσης να χαρακτηρίζονται από υψηλό επαγγελματισμό και καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση και στην κατάρτιση ε, των ενδιαφερομένων. Πιστεύω ότι με συνεργασία θα καταλήξουμε σε ισορροπημένη λύση προκειμένου η εσωτερική αγορά να είναι ολοκληρωμένη και ισορροπημένη και να ευνοεί ταυτόχρονα τους επιχειρηματίες, ε, τους πολίτες, τους καταναλωτές και σε τελική ανάλυση όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλντε, κύριε Κρότσιμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ε, παρουσίαση και για την ε, πρωτοβουλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι εφβέβαιος ότι θα αποβεί όφελο και θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον καταναλωτή και και τις μικρέ επιχειρήσει Μπορεί να συμβάλλει και στην ε, μείωση του κόστου και στην καλύτερη διαλειτουργικότητα και σε μια καλύτερη ε, κινητικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ωστόσο ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σχετικά νεαρό και πρέπει να το αφήσουμε το χρόνο για να αναπτύξει τις καλύτερες υπηρεσίες οι πιο ελκυστικές προσφορές είναι αυτές που θα πρέπει να αφήσουμε να ε, επικρατήσουν χάρη στην ποιότητά τους και να μην επιβάλλουμε με πρώιμη παρέμβαση λύσεις οι οποίες δεν θα ε, προστατεύουν τις αρχές της ε, καλής εσωτερικής αγοράς. Αλλά βλέπω ότι και ο εισηγητής αυτό επιδιώκει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλεί για μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών εκεί όπου είναι χρήσιμη, εκεί που μπορεί να προσφέρει προσθέμενη αξία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ειδικά όσον αφορά την, καταγραφή της, την αναγραφή της διεύθυνσης και την σήμανση του δέματος. Ο Η οδηγία για τον καταναλωτή μπορεί να έχει πιστεύουμε στην πρόταση αυτή τη δική της ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφέρεται και σε ελάχιστες ε, προθεσμίες για την ε, επιστροφή προϊόντων για το δικαίωμα ανάκλησης της ε, παραγγελίας και το καθεξής και, μπορεί να... και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παραπομπή κυρίες και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων και μπορούμε με το σύστημα αυτό να εξασφαλίσουμε απλούστευση των σχέσεων μεταξύ πολιτή και αγοραστή και να μην κινδυνεύουμε να αποτρέψουμε τον αγοραστή από την ενδεχόμενη επιστροφή ενός δέματος λόγω περίπλοκων ε, κανόνων ως προς την αναγραφή της διευθύνσεως. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό πιστεύω, θα ήταν καλό να το εξετάσουμε. Εν γέννη είναι πολύ λογική και ισορροπημένη η πρόταση του κύριου Αρίας και δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η πράσινη τώρα, η κυρία Ρούλε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι μια πολύ καλά σταθμισμένη έκθεση. Δεν μπόρεσα δυστυχώ να παραστώ στι συνεδρίε των σκιωδών. Αυτό δεν, δεν πρέπει να ε, σα δώσω την εντύπωση ότι δεν ε, βρίσκουμε καλή την έκθεση της σας των αντίον, τη θεωρούμε καλή και δεν βρίσκουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, βλέπουμε ότι έχετε δώσει μια γενική εικόνα για το τι θέλετε να καταγράψετε στην έκθεση. Θα ήθελα για το θέμα όμως του δικαίου των πωλήσεων να απαντήσω στον κύριο Κρόιτσμαν ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για την μοίρα που θα έχει όταν φτάσει στο Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μην πέσει μέσα σε αυτό το το πιθάρι με τις προτάσεις που δεν εγκρίνει το Συμβούλιο και ίσως θα ήταν καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην ενσωματώσουμε και άλλο θέμα το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο πολλές δυσκολίες στη σχέση μας με το Συμβούλιο. Η έκθεση είναι πολύ καλή. Έχει υπογραμμίσει τα σημεία σωστά και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλη κυρία Πιετικά, είναι κύριος Μπίλαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης. Είναι πολύ αξιόλογη έκθεση, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και χαίρομαι που προωθείτε το ηλεκτρονικό εμπόριο στηρίζοντας την αρχή της ελεύθερης αγοράς και όχι ε, κατάχρηση των ε, νομοθετικών επιβαρύνσεων ε, που ουσιαστικά επιβραδύνουν την ανάπτυξη του κλάδου. Θεωρώ ότι οι νέες νομοθετικές διατάξεις, αν υποβληθούν, να είναι πραγματικά αναγκαίες. Θα πρέπει να αποδειχθεί κάτι τέτοιο και κυρίως να αφήσουμε τον ίδιο τον κλάδο να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς. Ε, στο σημείο 16 μιλούμε για το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την οδηγία 83 του 2011 και την ανάγκη ε, υιοθέτηση αυτών των νομοθετικών διατάξεων μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Γιατί στο έγγραφο αυτό υπάρχουν πολλές ε, σημαντικές ε, οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για παράδειγμα το στερεότυπο έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης. Είναι σημαντικό επίσης να υποβάλουμε συστάσεις, αλλά να μην επιβάλλουμε στον κλάδο ε, ρυθμιστικά ή κανονιστικά μέτρα. Συμφωνώ λοιπόν με την σχετική τοποθέτηση του εισηγητού. Τέτοιες συστάσεις θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η, η συγκέντρωση των προσπαθειών για την βελτίωση των υπηρεσιών, ε, καλύτερη χρησιμοποίηση των μεταφορών για να μην έχουμε κενές ε, μεταφορές, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την μεγαλύτερη πρόσβαση των, ε, ε, την πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες, ιδιαίτερα για το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο και ε, αποφυγή της υπερβολικής επιβάρυνσης των επιχειρηματιών. Θεωρώ ότι θα βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ της ενημέρωσης και της υποχρέωσης των επιχειρηματιών στην σχετική οδηγία που έχουμε για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Είναι σημαντική η σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να διευκολύνουμε την, τις ε, συναλλαγές μέσω διαδικτύου και προβλέποντας κάποιες διατάξεις σχετικά με τη χρήση του κατάλληλου συναλλάγματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες καταβολής σε άλλο συνάλλαγμα από αυτό της, του καταναλωτή ή του επιχειρηματία. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα συγκριτικού πίνακα των τιμών για να διευκολύνεται ο καταναλωτής να διαλέγει τις πιο ευνοϊκές τιμές ε, όντας σε θέση να συγκρίνει τις τιμές παράδοσης. Πάντως, επαναλαμβάνω, η έκθεση βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση θα υποβάλω εδώ κάποιες τροπολογίες, αλλά ήδη από τώρα μπορώ να σας αναγγείλω ότι δεν θα απάδουν από τη βασική κατεύθυνση του εισηγητού μας. Ευχαριστώ. Thank you. And, uh... Δεν βλέπω άλλον σκιώδη συγητή. Ας ακούσουμε τους λοιπούς συναδέλφους. Κύριε Κορεία Κάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Παύλο Αρίας για μία ακόμη σημαντική έκθεση που ακολουθεί την παράδοση των ποιοτικών προηγούμενων εκθέσεων του. Από, τους πέντε, από τις πέντε βασικές μέρημνες των καταναλωτών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το θέμα της ποιότητας της παράδοσης είναι από τις πιο σημαντικές ανησυχίες. Και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ε, συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες επιφυλάξεις ε, λόγω των προβλημάτων παράδοσης που υπάρχουν. Ε, και προβλήματα δημιουργούν όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά στις επιχειρήσεις, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. σίγουρα είναι πολύ μικρότερη η αγορά μέσω διαδικτύου από ότι η αγορά στην εσωτερική αγορά. Αυτό δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και την απροθυμία τους να αγοράσουν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Άλλωστε μερικές φορές τιμές παράδοση είναι τόσο αστρονομικές ε, ακόμη και όταν ε, είναι πολύ κοντά ο προμηθευτής ε, με τον καταναλωτή μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται σε διαφορετική χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα αποτελεσματικό, διαφανές, αξιόπιστο σύστημα υπηρεσιών παράδοσης που θα εξυπηρετεί ε, σε το χρόνο και τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Έχουμε μια καλή αγορά και αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί μόνο τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Αλλά εμείς δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει κυρίως να μεριμνούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σωστό ο στόχος ε, του εισηγητού. Καινοτομία. Η καινοτομία σίγουρα ε, θα πρέπει να στραφεί στην προσαρμογή των ωραρίων, στην, ε, στην εγκατάσταση σημείων παραλαβής, στην, ε, στον εντοπισμό και παρακολούθηση του δέματος από την αρχή μέχρι την στιγμή της παραλαβής, όπου και αν είναι το σημείο παραλαβής και φυσικά να ευνοείται η παραλαβή ακόμη και στις απομονωμένες και απόμακρες περιοχές. Καλό θα ήταν να έχουμε και συγκριτικούς πίνακες των ε, ε, ισχυών των συστημάτων παράδοσης, γιατί υπάρχουν πολλά και διάφορα συστήματα παράδοσης αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πλούσιο παγκόσμιο εμπόριο, γι' αυτό και είναι χρήσιμο να κάνουμε μια προσπάθεια σύγκρισης ε, των διαφόρων ιστοσελίδων για να δούμε πόσο στοιχίζουν οι υπηρεσίες παράδοσης, τι προθεσμίες χρησιμοποιούν, ώστε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην ε, εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αρίας γιατί είναι πολύ καλή και ισορροπημένη η έκθεσή του και με τις ε, τροπολογίες που φαντάζομαι θα δεχτεί και ο εισηγητής θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος ομιλητής υπάρχει. Τότε παρακαλώ την Επιτροπή. και τον τμήματάρχη της ε, μονάδας ε3 της Γενικής Διεθνής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους όσοι έλεγαν τον λόγο και ιδιαίτερα τον εισηγητή για την πολύ καλή του έκθεση, αλλά και όλους και τους εισηγητές για την συμμετοχή τους και την πολύ καλή συνεργασία. Ε, καταγράφεται από τις σημερινέ ε, συζητήσεις συνένεση, την οποία βέβαια οφείλουμε στην πολύ ισορροπημένη διατύπωση της εκθέσεως του Παύλου. Αυτό μπορούμε να πούμε από πλευράς μας είναι ότι είναι πολύ θετικό το ότι το Κοινοβούλιο επισημαίνει τα ίδια προβλήματα και ζητήματα που είχαμε επισημάνει και εμείς ε, αλλά και δίνει τις ε, αντίστοιχες κατευθύνσεις ως προς το πώς θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Το να παρέμβουμε υπερβολικά ρυθμιστικά στο στάδιο αυτό, συμφωνούμε ότι θα ήταν υπερβολικό. Χρειάζεται ωστόσο να έχουμε ένα ε, πλαίσιο ευρύ, το οποίο θα παρακολουθούμε όμως στενά. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μέσα και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος, θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Αν όχι, ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον εισηγητή, τους συναδέλφους για τη συμμετοχή στο σύστημα, στο, στη συζήτηση. Έχουμε πει λοιπόν ότι 4 και 5 Νοεμβρίου θα συστηθούν οι τροπολογίες, ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπουμε. Κατάθεση τροπολογιών, διορθώνω, λέει η ομιλήτρια. 8 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι, εξέταση τροπολογιών 4 και ή 5 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση, ψηφοφορία στην Επιτροπή 16-17 Δεκεμβρίου. Κλείνω το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. To the next uh, point of the agenda. Και πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων και εποπτεία της αγοράς προϊόντων μαζί, τα σημεία 13 και 14 της τη διάταξη. Έχουμε συμφωνήσει να γίνουν οι τοποθετήσει από, τους, από τις δύο εκθέσεις στην αρχή και μετά να ακούσουμε τους και οδησηγητές και λοιπούς συναδέλφους και εκπρόσωπο της Επιτροπής για τα σχόλια. Γιατί είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους δύο εκθέσεις η κυρία Σουάλτε Μόζερ είναι καθοδόν. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, μια και έχω εγώ αναλάβει την εποπτεία της αγοράς, μπορώ να ξεκινήσω με την παρουσίαση. Έτσι μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο και να συνεχίσουμε με την παρατηρήση της κυρίας, με Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδες συζητητές για την πολύ επικοδομητική τους ε, προσέγγιση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κοινέ συνεδριάσεις με δύο εισηγητές ε, των δύο φακέλων αυτό και τους σκιώδεις. Ιδιαίτερα λοιπόν ε, επικοδομητικές συζητήσεις και ήδη τώρα εξετάζουμε τις τροπολογίες και μετά από αυτή την συνεδρία της Επιτροπής μας θα προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε τη βάση συμβασμού για να υπάρξει και ομοφωνία επί της ουσίας, όσο γίνεται βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, για να σας παρουσιάσω συντομία τις τροπολογίες σε αυτή την έκθεση για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων, μπορώ να πω ότι Η πλειονότητα των τροπολογιών αφορά τέσσερα σημεία. Τους ορισμούς, με τις ε, επιγραμμικές πωλήσει, μετά κυρώσεις, υποχρεώσεις οικονομικών φορέων εμπορευομένων και τρίτων μερών και αυτό συνδέεται με τους ορισμούς. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του νητρώου Για τους ορισμούς λοιπόν, η συζήτηση με εισηγητή συνεισηγητές σκιώδης ουσιαστικά αφορά το κατά πόσο υπάρχει, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον, ε, στην ασφάλεια και στον ε, ρυθμιστικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, από τροπολογίες SWAB και το καθεξής ε, αφορούσαν την ε, πρόταση διαφοροποίησης με τα προϊόντα που ε, δημιουργούν κίνδυνο για την ασφάλεια και κίνδυνο κανονιστικό. Η έννοια του κινδύνου ε, εμπεριέχεται εδώ γιατί έχουμε λάβει υπόψη και τιμή συμμόρφωση των προϊόντων. και μου φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ του κινδύνου για την ασφάλεια που μπορεί να προκαλέσει ε, κάποια ζημιά σε ό,τι αφορά την υγεία του καταναλωτή και την άλλη έχουμε και κινδύνους ε, μη συμμόρφωσης. Μια ενδεχόμενη λύση θα ήταν μια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο, αντί όμως, αλλά να μην έχουμε πραγματικό διαχωρισμό μεταξύ των δύο έτσι να έχουμε λοιπόν μια δυνατότητα να πάμε παραπέρα, να ε, εντοπίζουμε διαφορετικούς ε, τύπους ε, κινδύνου ή να το εντάξουμε αυτό στους ορισμούς, ούτως ώστε να έχουμε αφενός τους κινδύνους και αφετέρου μια ξεκάθαρη κατηγορία μη συμμόρφωσης. Τώρα, τα προϊόντα που παρουσιάζουν αναδεόμενο κίνδυνο. Είναι και αυτό ένα θέμα στους ορισμούς. Κάποιες ε, τροπολογίες ε, προτείνουν ε, τέτοιοι κίνδυνοι αφορούν μόνο τα μη εναρμονισμένα προϊόντα. Τα μη εναρμονισμένα θα καλύπτονται από αυτό γιατί η εναρμόνιση καλύπτει έτσι καλλιώς ε, τον κινδύνο και δημιουργεί αυτομάτως την ασφάλεια. Όμως, εξορισμού, ο αναδυόμενος κίνδυνος είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε το οποίο την ύπαρξη ακόμα δεν γνωρίζουμε και έτσι ε, δυσκολευόμαστε να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων. Γιατί πρόκειται για κινδύνους που δεν τους γνωρίζαμε. Όταν ε, προετοιμάζαμε τον κανονισμό για τα αναρμονισμένα και αναρμονισμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, ε, έχουμε στην περίπτωση των παιχνιδιών ε, κάποιες περιπτώσεις όπου δεν ήταν γνωστός ο κίνδυνος και δεν είχε τύχει ρύθμισης στην οδηγία, αλλά όπου ήταν απαραίτητη η απαγόρευση. Όταν εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό και μου φαίνεται δύσκολο να κάνω μια, μια τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων σε ό,τι αφορά τους ε, αναδυόμενους κινδύνους. Μετά, οι διαδικτυακές πωλήσει. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις που αφορούν το σημείο αυτό, τον πωλήσεων στο διαδίκτυο, σε διάφορα σημεία του κανονισμού. Ο σκοπός του κανονισμού είναι να καλύψει και τις ε, πωλήσει στο διαδίκτυο και τις άλλες μορφές πωλήσεων. Ίσως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση, ούτως ώστε να, να προτείνουμε ένα εκτιμώντας που να υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του κανονισμού και ότι σκοπός είναι να καλύπτονται και οι δύο μορφές πολίσεων, και στο διαδίκτυο και εκτός. Αυτό υπάρχει και σε προηγούμενες οδηγίες, επομένω ε, σίγουρα θα βρούμε μια καλή λύση. Οι κυρώσεις τώρα είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε εκτενώς. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υψηλές, αυστηρές οι κυρώσεις. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι το σημείο αυτό για τις κυρώσεις αφορά την εισαγωγή κινδύνων, τη σκόπιμη εισαγωγή ε, κινδύνων και μη Δεν ε, μιλάμε για μια περίπτωση όπου κατά λάθο κάποιος έβαλε ένα άλλο ε, εμπορικό σήμα ή όταν κατά λάθο προκύπτει ένας θάνατος ανθρώπου παρότι ο αρμόδιος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Εδώ σκοπός μας είναι η αποτροπή και θέλουμε να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τη διατύπωση ε, της νομοθεσίας αντιτράστη της Ένωσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και δεν θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στις αγορές μας ε, κάποιος ε, σκοπίμος να βλάψει τους ε, καταναλωτές και να προσπαθήσει να αποφεληθεί. Ελπίζω να υπάρξει συμφωνία σε ό,τι αφορά τις ε, κυρώσεις, όταν μιλάμε για την σκόπιμη εισαγωγή κινδύνου από τα προϊόντα. Μετά υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις και συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι φορά τις υποχρεώσει των εμπορευμένων. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε πιο επισταμένα αυτό το πιο τεχνικό ζήτημα για να ευθυγραμμίζονται όλοι οι κανονισμοί είτε μιλάμε για την υποπτήρια της αγοράς είτε τη συμμόρφωση των προϊόντων. Υπάρχουν ακόμα κάποιες υποχρεώσεις που θα πρέπει να προσθεθούν εδώ. Θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε το τμήμα που αφορά την εποπτεία της αγοράς όπως οι διατάξεις για την υποχρέωση για τους κατασκευαστές που ε, εδράζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονοματίσουν έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκρινίζουν ε, τη σειρά με την οποία ε, κοινοποιείται η απαραίτητη τεκμηρίωση της αρχές. Αλλά έχουμε καταλήξει σε συμφωνία προς αυτό. Τέλος, συζήτηση για το RAPACS αν θα πρέπει να αφορά τους σοβαρούς κινδύνους ή όλους τους κινδύνους. Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ακούω διαφόρους εμπειρογνώμονες που έχουν διαφορετικές απόψεις. Αφενός είναι σωστό ότι ε, θα πρέπει να αφορά μόνο τους σοβαρούς κινδύνους και να μην ε, αναλωνόμαστε με όλα τα μικρά τεχνικά ζητήματα. Από την άλλη όμως, το να έχουμε πολλές παρατηρήσεις και από την Επιτροπή, αλλά και από τις αρχές εποπτείας ε, στα επιμέρους κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, τέτοια ποικιλομορφία στις ερμηνείες του κάθε κράτους μέλους και της κάθε αρχής για το τι σημαίνει σοβαρός κίνδυνος, που βλέπουμε ότι ακόμα και την ίδια ημέρα, την ίδια εβδομάδα, ε, έχουμε διαφορετικές κατεχωρήσεις ε, του ίδιου περιστατικού. Σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται ως σοβαρό περιστατικό και σοβαρός κίνδυνος και σε άλλες ως απλός κίνδυνος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αναδυόμενους κινδύνους. Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος υπάρχει, κίνδυνος υπάρχει για παράδειγμα, ε, κάτι το οποίο μπορεί να μην ε, σκοτώσει κανέναν, για παράδειγμα, απευθεία, αλλά να έχει πολύ σοβαρέ ε, ε ρηπαντικέ ουσίε ένα ρούχο, για παράδειγμα. Και έτσι ίσως θα ήταν καλό να έχουμε όλους τους κινδύνους μέσα από το Μητρό. Από την άλλη υπάρχει διαφορετική άποψη ότι θα μπορούσαμε να απαλείψουμε τις ίσονος σημασίας κοινοποιήσεις Ίσως μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα και πάλι στους ορισμούς και να μιλάμε μόνο για ρυθμιστικό, κανονιστικό κίνδυνο ή να έχουμε ξεχωριστή κατηγορία μη συμμόρφωσης. Θέλω όμως να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να φορτώσουμε το μητρό με όλες τις ε, δευτερεύουσες λεπτομέρειες, αλλά ούτε απ' την άλλη για να χάσουμε και το, τα επίπεδα ασφαλείας που θέλουμε από αυτό το μητρό, γιατί διαφέρουν οι ερμηνείες ανάμεσα στα κρατημέλη. Καλό ήταν, θα ήταν λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Στρέφομαι τώρα προς εσάς, ε, να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις πριν ε, δώσουμε το λόγο στους Χιώδης, ε, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για την ε, ασφάλεια προϊόντων. Ξεκίνησα νωρίτερα γιατί είχαμε χρόνο και ήξερα ότι θα φτάσει σε λίγο. Γι' αυτό ξεκίνησα με το επόμενο θέμα. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. θα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, με μία ψηφοφορία για τον ε, ιατρικό ε, εξοπλισμό και πρέπει να σας πω ότι πολλές από τις δικές μας ε, τροβολογίες από τη γνωμοδότηση έγιναν δεκτές. Τώρα τι θέλετε, θέλετε να κάνω μια παρουσίαση του δικού μου τμήματος και να σχολιάσω και το δικό σου. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το καταλληλότερο. Πρώτα να κάνεις το δικό σου, να παρουσιάσεις τη δική σου έκθεση και μετά ως σκιώδης και αλλάζοντας ε, καρτελάκι να αναλάβεις να σχολιάσει το δικό μου τη δική μου έκθεση. Καλώς. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ όλους τους και ηγητές για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Έδειξαν πολύ καλή διάθεση και προσπάθεια για τη σύνταξη μιας καλής έκθεσης. Αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε, καταρχάς μπορούμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές λύσεις και ταυτόχρονα πιστεύω θα μπορέσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το νομοθέτημα πριν το πέρα της ε, θητείας μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα εκθέσω κάθε στοιχείο της εκθέσεως μου. Θα προσπαθήσω απλώς να σας παρουσιάσω τους τομείς τους οποίους θεωρώ πιθανό και επιθυμητό να προχωρήσουμε σε συμβαστικές ε, λύσεις. Εννέα είναι οι τομείς τους οποίους μπορούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Έχουμε καταρχάς συζήτηση για το πεδίο και την ασφάλεια των προϊόντων σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες και εδώ θα πρέπει πιστεύω να βρούμε συμβαστικές λύσεις γιατί είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε στο πώς θα ερμηνεύουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Άρα μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Επίσης ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για τους ορισμούς για προϊόντα απευθυνόμενα στα παιδιά τα οποία μιμούνται την εμφάνιση των τροφίμων. Και θα πρέπει να έχουμε μια κατηγορία κυρώσεων σαφή, ώστε να μην ε, τολμάει κανείς να παραβεί την ομοθεσία, να, να, δρά πραγματικά αποτρεπτικά. Και εκεί θα έλεγα με μέλημα πάντα την ε, ασφάλεια του καταναλωτή και όχι τόσο το να τιμωρηθεί η παραβίαση, η μη, η μη συμμόρφωση. Για το σήμα CE, Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ε, ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Αγορά. Ξέρουμε και συμφωνείτε πιστεύω περισσότεροι ότι είναι ένα σήμα το οποίο πλέον μπορεί να ε, θεωρείται έως παραπλανητικό για τον καταναλωτή και άρα θα συζητήσουμε πιστεύω ή το να εισαγάγουμε ένα νέο σήμα CE+, συν, ώστε να είναι πιο ασφαλές ή αλλιώς και να αποσύρουμε τελείως το σήμα C. Πάντως το βασικό είναι να έχουμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό κατά τρόπο ώστε να είναι χρήσιμος και απλός και κατανοητός για το καταναλωτή. Η απόσυρση της αναφοράς στην αρχή της πρόληψης την οποία ζητάει η Επιτροπή. Το έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται πραγματικά, γιατί και η Επιτροπή ξέρει πολύ καλά τι πιστεύω. Δεν συμφωνώ να αποσυρθεί η αρχή της πρόληψης. Αλλά δεν έχω καμιά αντίρρηση να το συζητήσουμε, να συζητήσουμε πάνω απ' όλα πού θέλουμε να ε, εγγράψουμε αυτήν την αρχή, σε ποιο σημείο του κειμένου. Επίσης, για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο κανονισμός αυτός. Θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, άρθρα 2, 5 και 6, τις προτάσεις στα οποία έχουν κατευθεί αρκετέ τροπολογίε, πιστεύω και νομίζω ότι μπορούμε να τις ε, συζητήσουμε και να βρούμε κοινού ορισμούς. Τροπολογίες πολλές έχω δει επίσης από πλευρά σας για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές και τις προβλέψιμες πιθανές ε, συνθήκες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα το συζητήσουμε και ιδιαίτερα για τους ευάλωτους καταναλωτές. Ε, πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει να έχουμε συναντήληψη στην υπόθεση αυτή. Και στο θέμα των οικονομικών φορέων νομίζω ότι η υποχρέωση την οποία, με την οποία επιβαρύνουμε τους οικονομικούς φορείς είναι τέτοια που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωσή μας και αν μπορέσουμε θα ήθελα χωρίς να ανατρέψουμε τα όρια της ευθύνης σε όλη αυτή τη διαδικασία της αλυσίδας προμήθειας να καταστήσουμε, να καταφέρουμε να καταστήσουμε σαφές και κατανοητό αυτό που ζητάμε από τον οικονομικό φορέα. Αλλά να μπορούμε να έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό βέβαια για το θέμα αυτό. Με όλη αυτή δέσμη. Και αντίστοιχα βέβαια αποτελέσματα με αυτά τα, τις εποπτείες της αγοράς προϊόντων. Ε, σε σχέση δε με το άρθρο 13 και την αποδοχή κάποιων ε, κανόνων για τους οικονομικούς ε, φορείς. Ε, χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον με επιπλέον επιβάρει με επιπλέον φόρτο ή κόστος, ε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις που να τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη διαθέση αγορά. Για το άρθρο 7 όμως, και ξέρω ότι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές ήδη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε συμβασμό στην υπόθεση αυτή για την ε, ε, προέλευση, του κανόνε προέλευση. Είμαι υπέρ τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε όμω να βρούμε συμβαστικέ λύσει. Πιστεύω και προτιμώ να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και να καταλήξουμε με την ψηφοφορία για το αν θα υποστηρίξουμε τι θέσει τη Επιτροπή, τι οποίε θα υποστηρίζω εγώ για την ένδειξη καταγωγής ή προελεύσεως. Άλλα θέματα στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε υπάρχουν. Αλλά εγώ σε αυτά ήθελα να επικεντρωθώ και σε αυτά σκοπεύω να ε, συγκεντρώσω το ενδιαφέρον μου για τις συμβαστικές τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια αναγορά εσωτερική για τα προϊόντα, για τα τεχνολογικά προϊόντα. Ε, το χρονοδιάγραμμα μας έχει απασχολήσει επίσης σε συζητήσεις των ε, σχεδόν εισηγητών και των συντονιστών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή και της ενδεχόμενη έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη συνένεση, είμαι διτεθειμένη να ε, προβλέψω συμπληρωματικές συναντήσεις με τους κοιόδης συγητές, χωρίς όμως να αλλάξω την τελική ημερομηνία για την ψηφοφορία. Θα απλώς θα φροντίσω ενδιαμέσως να οργανώσω συναντήσεις για να ξανασυστήσουμε οποιοδήποτε θέμα θα ήταν πρόσφερο για συμβασμό. Ένα-δύο λόγια τώρα για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους οι ορισμοί στα δύο αυτά νομοθετήματα. Αλλά πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό, γιατί αν συμφωνήσουμε σε έναν ορισμό, αυτομάτως ε, τον ενσωματώνουμε στην, ε, στον ορισμό στη μία έκθεση, αυτομάτως τον ενσωματώνουμε στην άλλη ή μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία μια συμβουλή για το που είναι το καταλληλότερο σημείο για να καταγραφούν οι ορισμοί. Ρέιπεξ, και συμφωνώ μαζί σου, ότι το το η Rapex θα είναι ίσως δύσκολο να το λύσουμε. Έστω, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε ή να διακρίνουμε την περίπτωση της μη τήρησης ή της μη ε, συμμόρφωσης από τον κίνδυνο. Γιατί άλλο είναι το να μη συμμορφούνται ο ε, ο κατασκευαστής και άλλο να προξενεί κίνδυνο και όταν βλέπει το όνομά του σε κάποια βάση η οποία έχει να κάνει με την καταγγελία της μη συμμόρφωσης φαντάζομαι ότι θα κάνει μια προσπάθεια παραπάνω για να μην μπαίνει το όνομά του σε αυτό. Αλλά να έχουμε έναν εσωτερικό δίκτυ στο RAPEX, έναν, ε, ε, έναν κατάλογο περισσότερο ο οποίος θα αφορά μόνο τον κίνδυνο και έναν άλλο κατάλογο ο οποίος θα καταγράφει την μη συμμόρφωση, ώστε να διακρίνεται αυτή από τους σοβαρούς κινδύνους. Επίσης, τα κράτη-μέλη πιστεύω θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους, πιο σοβαρή ε, δηλαδή δραστηριοποίηση για την ε, εποπτεία της αγοράς προϊόντων. Πολλά ακόμα μπορούν να κάνουν και πρέπει να κάνουν. έχω και κάποιες ιδέες για ελάχιστες προδιαγραφές για την επαλήθευση προϊόντων ε, που διατίθεται στην αγορά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο 0,3% των προϊόντων που δείχνεται στην αγορά ε, ελέγχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα ελάχιστο ποσοστό στο 2% φερρυπίν. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε, αλλά πάντως πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη και να τα πιέσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους προς την εποπτεία της αγοράς. Καταθέτω επίσης Προτάσει για την ε, πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων ε, και στο δικό μου κείμενο και στο δικό σου. Είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη και εστιασμένη ε, νομοθεσία ώστε να εντοπίζουμε γέρο τα πραγματικά επικίνδυνα προϊόντα. Κυρία Πιέτικα, δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές στις δύο εκθέσεις. Είμαστε σχεδόν στην ίδια γραμμή. Και επιδιώκουμε και οι δύο την, τον ίδιο στόχο, δηλαδή μια πιο αποτελεσματική εποπτεία στις αγορές που δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα κοιτάξουμε βεβαίως τώρα, θα ακούσουμε μάλλον τις απόψεις των ε, σκιωδών εισηγητών, ε, της ε, κυρίας Άλτερ Μόζερ, καταρχάς ο κύριος Μπαλτασάρε νομίζω ήταν. Α, ήταν εδώ πριν από λίγο, νάτος. Ξεκινώ μαζί σας, κύριε Μπαλτασάρε. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Κρόιτσμαν, ο οποίος έχει αναλάβει και τις δύο εκθέσεις. Όχι, ο κύριος Χέλβικ έχει αναλάβει την άλλη. Μία εγώ, μία ο κύριος Χέλβικ. Καλώς και κυρία Ρούλε μετά τέταρτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και την Πρόεδρο, κυρία Πιτικάιναν, για το έργο της και τη συνεργασία της με τους ε, σκιώδεις. Δεν χρειάζεται να μείνουμε για πολλή ώρα σε αυτές τις δύο εκθέσεις, γιατί ήδη έχουμε κάνει τις συζητήσεις. Το θέμα είναι μόνο να εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και ενδεχομένως να δώσουμε και τις δικές μας απόψεις ε, επί των τροπολογιών. Και εγώ κατέθεσα τροπολογίες επί του πεδίου εφαρμογής γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερο να εξηγήσουμε ποια προϊόντα αφορούν τους καταναλωτές, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν λιγότερες δυσκολίες και μεγαλύτερη σαφήνεια. Τώρα στο άρθρο 3 και τον ορισμό του ασφαλούς προϊόντος θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να ευθυγραμμιζόμαστε με τα πρότυπα εναρμόνισης ε, ασφάλειας και υγείας με τα αντίστοιχα πρότυπα. Στα, στο άρθρο 6 για την αξιολόγηση της ασφάλειας υπάρχει ένα σύνολο κριτηρίων που ισχύουν και εφαρμόζονται όταν υπάρχει έλλειψη ορισμού σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, την τεχνολογία εχμής, την ασφάλεια του καταναλωτή, ασφάλεια που προσδοκά ο καταναλωτής, άρθρο 6, παράγραφος 2. Νομίζω ότι αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και διαθέσιμα στους ε, κατασκευαστές. Τεχνολογία εχμής και οι ε, θεμητές και θεμητές ε, προσδοκίες του καταναλωτή επιδέχονται διαφόρων ερμηνεών από τους καταναλωτές, ή ε, από τους κατασκευαστές, συγγνώμη. Μετά, άρθρο 8, ε, η υποχρέωση διατήρησης των εγγράφων για 10 χρόνια, ίσως είναι λίγο περιβολικό, αλλά είναι καλή ιδέα να είναι διαθέσιμα, αλλά ίσως όχι για 10 χρόνια. Και μετά η υποχρέωση του διανομέα δεν μπορεί να, είναι, να διασφαλίζει ότι ε, συμμορφούνται οι εισαγωγείς με τους κανόνες δεν είναι δική τους αρμοδιότητα αυτή. Εκείνοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι το προϊόν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν τη συμμόρφωση. Τώρα, υπάρχουν υποχρεώσεις που ανέφερε η συγγήτρια, το θέμα των εμπορευομένων. Στο κεφάλαιο υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις για τους εμπορευομένους οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες σε αυτό το κεφάλαιο και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να επικεντρωθούμε στο κείμενο που υιοθετήθηκε χωρίς να επιφέρουμε περαιτέρω αλλαγές στο δίκτυο ασφαλείας η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να είναι η μόνη νομοθετική πράξη που θα πρέπει να ε, σέβονται και να τηρούν ε, οι κατασκευαστές. Τώρα, για τα σήματα, το marking, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες που μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε ε, αβεβαιότητα όταν έχουμε πολλά σήματα τέτοια CE+. Ε, με σπατάλη χρόνου και οικονομικών πόρων, αλλά και με πολύ μεγάλο άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την αρχή της αναλογικότητας τώρα θα ήθελα να επαναλάβω τις ε, επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί. Τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μπορεί να οδηγηθούμε και πάλι στην ε, νομική αβεβαιότητα. Ε, η αρχή αυτή ε, συμπεριλαμβάνεται στον ε, ορισμό του ασφαλούς προϊόντος που μιλά για προβλέψιμες χρήσεις. Τώρα για τις κυρώσεις όταν υπάρχει παράβαση των κανόνων ασφαλείας έχουμε τον ορισμό CPR και MSR. Ίσως ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, ορισμός ε, για τις κυρώσεις και ίσως είναι ο κανονισμός για την εποπτεία των αγορών που θα πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες. η τροπολογία του κ. Κρότσμαν είναι μια καλή πρόταση. Τώρα, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμφωνώ πράγματι είχε συζητηθεί επί μακρόν. Ξέρω ότι ο κύριος Κρόιτσμαν ε, ε, ταράσεται όταν το συζητούμε, αλλά δεν είναι και ταμπού. Στην Γιούρη, στην Ίντα, ακόμα ίσως και στην Ήτρε υπήρξε πολύ μεγάλη πλειοψηφία ως προς αυτή τη θέση και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των ε, ζητημάτων που αφορούν τις, αγορές, τις αρχές εποπτείας της αγοράς και της ε, διαθεσιμότητας πληροφοριών στους ε, καταναλωτές για τα περίοδα που αγοράζουν. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το γεγονός ότι ένα, από τα 10 προϊόντα, ένα στα 10 προϊόντα είναι μη ασφαλές ε, και δεν έχει γεωγραφική ένδειξη προέλευσης. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε που επιβάλλουν γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης στις ε, χώρες που εξάγουν προς τη δική τους χώρα. Επομένως, δεν αφορά μόνο την αύξηση της ασφάλειας του προϊόντος, αλλά και της διασφάλισης της αμοιβαιότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών εταίρων της. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική του προσπάθεια και το εξαιρετικό του έργο. Νομίζω ότι πολλές ε, επιτροπές έχουν καταφέρει να καταλήξουν συμφωνία από αυτού και νομίζω ότι και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπαλτασάρε. Και περνάμε στην άλλη. Κύριε Κρόιτσμαν, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Χέλβικ, νέος συνάδελφος στο Κοινοβούλιο, θα αναλάβει να μιλήσει για την εποπτεία ε, και τι πολλές από τις τροπολογίες έχουμε συντάξει μαζί. Εγώ επικεντρώνομαι λοιπόν μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των ε, ε, διατάξεων για εναρμονισμένα και μη εναρμονισμένα προϊόντα. Δεν μπορεί να μιλάει για εναρμονισμένα προϊόντα η οδηγία για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, τη σύμπτωση δηλαδή διατάξεων με άλλα νομοθετήματα. Τα, οποία, τα θέματα αυτά ήδη καλύπτονται από άλλες νομοθεσίες, λοιπόν από άλλες οδηγίες και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων καταναλωτικών προϊόντων. Ε, άλλο είναι τι είδου διατυπώσεις ή προϋποθέσεις ορίζουμε για, τους, ε, για, για την επιχείρηση και τι επιβάρυνση μπορούμε να τις επιβάλλουμε και άλλο το πώς θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε μια καλή λειτουργία τη αγορά. Αγαπητέ φίλε Μπαλτασάρε, δεύτερον, η σήμανση. Η σήμανση έχει να κάνει με την ε, ε, μη υποχρεωτική δήλωση μιας προελεύσεως, που ως εκ τούτου βρίσκεται εκτός ενός νομικού πλαισίου και δεν μπορεί να προσφέρει προσθέμενη αξία για την ασφάλεια που μπορούμε να θέλουμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή ή για την ορατότητα που θέλουμε ενδεχομένω για τα προϊόντα διαφορετικά είναι τα πράγματα όσον αφορά τις εναρμονισμένες διατάξεις δικαίου, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες διατυπώσεις, παραδείγματι ε, καταγραφή ονόματος διευθύνσεως, ε, ε, εισαγωγέα ή κατασκευαστή και ούτε καθεξής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν πάνω απ' όλα με την προστασία του καταναλωτή. Οι οργανώσει λοιπόν για την προστασία των καταναλωτών με τις οποίες εγώ επικοινωνώ και σήμερα ακόμη μιλήσαμε σε μια διαφορετική εκδήλωση ε, τοποθετήθηκαν κατά αυτές τις προτάσεις. Και εν τέλει, και σας το λέω κυρία Σουάλτε Μόζερ ρητά, διαρκώς μιλάμε για την περιστολή της ε, γραφειοκρατίας, για να το πω διαφορετικά, Δευτέρες λέμε πολύ γραφειοκρατία να την περικόψουμε, Τρίτη ερχόμαστε με αυτές εδώ τις προτάσεις. Ε, δεν γίνεται λοιπόν. Γιατί μη μόνο ότι έχουμε να κάνουμε με ομίλους, με θηγατρικέ εταιρείε κτλ. οι οποίες ε, πολλές φορές δεν μπορούν να δώσουν καν την ορατότητα του ποιο έχει παραγάγει τι. Για να μην μιλήσω για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πάρει ένα κομμάτι από εδώ και ένα κομμάτι από εκεί και δεν είναι σε θέση να ε, δώσουν ε, απόγραφη. Ξέρω κύριε Μπαλντασάρη ότι εσείς έχετε το σήμα το Ιταλικό στην Ιταλία, ξέρω ότι και για ε, πολλούς άλλους είναι σημαντικό αυτό, αλλά εγώ θα επιμείνω και αν το σκεφτείτε καλά-καλά δεν προσφέρεται τίποτα ως προς την ασφάλεια των προϊόντων. Ίσως είναι διαφορετικές οι πολιτικές σταθμίσεις, αλλά εν πάση μπορεί να, βρεθούμε κάποια, να βρούμε κάποια λύση ή να επικρατήσει μια διαφορετική πλειοψηφία. Η έννοια τώρα του ευάλωτου καταναλωτή ή του προϊόντος που απευθύνεται σε παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πάλι με βάση τον κίνδυνο και με μέλημα την θέσπιση ορθολογικών διατάξεων δικαίου. Το... Η αρχή της προλήψεως, αγαπητοί συναδελφοί, caution principle. Στο... Όταν μιλάμε για περιβάλλον, έχει βέβαια τη σημασία της. Γιατί μας ενδιαφέρει η αηφορία και ούτω καθεξής. Αλλά για πείτε μου λίγο ο επιθεωρητής που θα βγει σε ένα χωράφι για να ασκήσει την εποπτεία αγοράς. Πώς θα ξέρετε ότι έχει τηρήσει την αρχή της προλήψεως. Πώς, πώς θα βεβαιωθεί ότι τηρείται η αρχή της προλήψεως σε μια επιθεώρηση από τον επιθεωρητή. Και πώς θα πει μετά αυτός επιθεωρητής ότι ναι, όχι μόνο έχουν ε, ε, παραβιαστεί οι κανόνες περί ασφάλειας των προϊόντων ή όποιοι άλλοι κανόνες του οποίους θα πρέπει να συμμαρφώνεται, αλλά και η αρχή της πρόληψης. Καλή σας τύχη αν τα καταφέρετε. Εμείς θα κλεντήσουμε στη Γερμανία άμα, το, άμα περάσει αυτό το θέμα. Επίσης δεν πρέπει να ρεοσμονούμε την ανάγκη να προστευθεί η βιομηχανική ιδιοκτησία και πάνω απ' όλα το βιομηχανικό απόρριτο ή το επαγγελματικό απόρριτο. Πρέπει επίσης όταν μιλούμε για μη εναρμονισμένα προϊόντα να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά την επιχείρηση και να μην επιβάλλουμε διατάξεις πιο αυστηρές από αυτές που ισχύουν για τα εναρμονισμένα προϊόντα. Η διάρκεια της διατήρησης των εγγράφων των 10 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον κύκλο των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων. Και κύριε Μπαλτασάρη, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σα. Πέντε χρόνια ίσω να ήταν μια λογική λύση, αλλά δέκα χρόνια μου φαίνεται παράλογο. Και μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο ε, παραγωγός να δίνει στοιχεία είτε με το προϊόν μέσα στη συσκευασία είτε στην στον, ιστό στον του ενδεχομένως και με τη μορφή ακόμη απεικονίσεων, pictogram, για να ενημερώνει ε, ε, ικανοποιητικά τον καταναλωτή. Η προστασία του απορρίτου ή του μυστικού. Δεν πρέπει να υπάρχει ο κίνδυνος με την υποχρεωτική αυτή αναφορά των στοιχείων παρασκευής του προϊόντος να εκτίθεται στην απομίμηση και την υποβάθμιση της αξίας του προϊόντος του ο παραγωγός σε περίπτωση που κάποιος ε, από τρίτη χώρα αντιγράψει ή απομιμηθεί το προϊόν του. Άρα λοιπόν η, τα στοιχεία θα πρέπει να αφορούν μόνο τα, κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης για τις αρχές ε, στα στοιχεία αυτά αλλά με διαφορετικό τρόπο. η ε, ακρίβεια των πληροφοριών που διαθέτει είτε ο κατασκευαστής είτε ο εισαγωγέας θα πρέπει να επαληθεύεται αλλά δεν μπορεί η επαληθεύουσα αρχή να κρίνεται υπεύθυνη για την ανακρίβεια αυτών των στοιχείων. Γιατί αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι να επιτρέψουμε σε όλους τους κατασκευαστές και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να, κάνουν, να προσαρμόζονται στις συνθήκες ε, της νομοθεσίας χωρίς περιττή επιβάρυνση. Για τα θέματα λοιπόν αυτά και έχοντας επικοινωνήσει και με εκπροσώπους ε, των καταναλωτών πρέπει να σας πω ότι ε, στην πρόταση για την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού σήματος SIN, CE+, έχουν να παρατηρήσουν το εξή, ότι δεν προσθέτει τίποτα περισσότερο σχέση με το CE. Το μόνο που κάνει αυτό το σήμα είναι να επιβαρύνει με περισσότερο κόστος και πάνω απ' όλα να δίνει μία να, να εισάγει την έννοια της πλάνης για τον καταναλωτή, σαν να του δίνουμε μια διαβεβαίωση ότι το προϊόν που έχει το σήμα CE+, είναι πιο ασφαλές από το σήμα CE. Ε, e. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο η πρόεδρο. Και τώρα, αν, δεν έχετε αντίρρηση, α ακούσουμε έναν άλλο σκιώδη για το ίδιο θέμα. Ο κύριο Χέλβικ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ε, για τα καλά σας λόγια στην αρχή της συνεδρίασης. Θα ήθελα να πω ότι παρότι παραμένουν μόνο ακόμα μερικοί μήνες ε, για τη θητεία μας, ελπίζω η δική μου συμβολή στα νομοθετικά κείμενα που προετοιμάζουμε εδώ θα είναι θετική. Εδώ πρόκειται για πράγματα που με απασχολούν ιδιαίτερα. Θα ήθελα βεβαίως να συμμετάσχω στην καλύτερη ε, λειτουργία της Επιτροπής μας και σε πιο εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την εποπτεία των αγορών, στηρίζω τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι κυρία Νικολάη και Κρότσμαν. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις μου για να επισημάνουμε ακριβώς αυτά που μας απασχολούν. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το γενικό σκοπό του κανονισμού, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι οι κανόνες που αφορούν την εποπτεία των αγορών θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, ομοιόμορφα, ανεξαρτήτως της αλυσίδας ε, διανομής που ακολουθείτε. Για παράδειγμα, οι υποχρεώσεις για τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών με τη συνεργασία με τις αρχές υποπτήρες αγορών. Εδώ αναφέρομαι στην διαδικτυακή πλατφόρμα για την εμπορευματοποίηση των προϊόντων. Μετά, για τις υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας, όπως και άλλοι θεωρώ και εγώ ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και στη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναρμόνισης. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι αρχές εποπτείας θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην ε, διαδικασία τυποποίησης. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της ε, νομοθεσίας θα εξαρτηθεί από ε, τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ξεκάθαρο καταμερισμό και σε ό,τι αφορά το ε, άρθρο 8 περιορίζει τον αριθμό των αγράφων που μπορεί να ζητήσουν οι εμπορευόμενοι. Είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί ο καθένας θα πρέπει να θέτει ε, και να διαθέτει τα έγγραφα που αφορούν το προϊόν που θέτει σε εμπορία. αυτή η διάθεση θα, θα πρέπει να αφορά χείμενα που μπορεί να είναι είτε στο ε, διαδίκτυο είτε ε, επί χάρτου. Μετά γίνεται αναφορά για τα προϊόντα που δεν ε, συμμορφούνται, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και απαραίτητο επικίνδυνα για τον καταναλωτή. Εκεί οι αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν αν υπάρχει λόγος να γίνει αξιολόγηση κινδύνου για αυτό το προϊόν. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου στο άρθρο 13 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια κοινή μεθοδολογία για το συντομότερο δυνατόν. Κοινή μεθοδολογία λοιπόν για όλα τα κρατημέλη και η Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια διαδικασία μέσω εφαρμοστικών πράξεων. Σε ό,τι αφορά ε, τα κριτήρια ασφάλειας, ε, τρία κριτήρια ακολουθούνται στις αξιολογήσεις κινδύνου. Δεν είναι φυσιολογικό όταν ε, ένα προϊόν τηρεί την ομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι αρχές να μπορούν ωστόσο να λαμβάνουν μέτρα επειδή υπάρχουν νέες αποδείξεις που έχουν εμφανιστεί εντωμεταξύ. Αυτό δεν στέκει από νομικής πλευράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, ε, την απαγόρευση ή το μπλοκάρισμα κάποιων ε, προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βρούμε μια λύση για να αποφύγουμε αυτή την, αυτό το μπλοκάρισμα προϊόντων. Για το σύστημα RAPEX, νομίζω ότι οι κοινοποιήσει μέσω του συστήματο RAPEX θα πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στα προϊόντα που παρουσιάζουν πολύ σημαντικό κίνδυνο. Εάν το σύστημα φορτωθεί με έναν υπερβολικό ρυθμό κοινοποιήσεων, τότε θα μειωθεί πολύ σημαντικά και η ικανότητα ανταπόκριση των κρατών μελών. Κλείνοντας, ε, θα αναφερθώ στις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31. Το σύστημα που προτείνει η ομάδα μου, το Φιλελευθέρων, ε, ε, έχει ως αφετηρία την ε, νομοθεσία αντιτράστα του δικαίου ανταγωνισμού. Πρέπει να έχουμε μια κοινή μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε ό,τι φορά την ε, σοβαρότητα, την διάρκεια ε, και το καθεξής. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ποσοστό της, επί της πώλησης του προϊόντος αυτό είναι πιο εξισορροπημένο από ότι η πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κείμενο. Βεβαίω και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για όλα αυτά τα θέματα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ε, του κανονισμού, για να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμό μα ε, στο τέλο θα είναι ένα εργαλείο ε, για την αποτελεσματική εποπτεία των αγορών. Ευχαριστώ. Thank you, then, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούιλα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη. Εν περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, παρισταμένου για την πολύ καλή συνεργασία. Βλέπω να δουλεύουμε σαν πολύ καλή ομάδα και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή και πιστική εργασία, ένα καλό και πιστικό αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε την υποστήριξη του Συμβουλίου για να εγκριθεί το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια τη θητεία μα, γιατί αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο και άρα θα πρέπει να δείξουμε και πόσο σημαντικό είναι το θέμα και πόσο μεγάλη ευελιξία μπορούμε να δείξουμε. Πάνω απ' όλα πρέπει να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να κλείσει το θέμα αυτό μέσα στη θητεία ε, και πρέπει να κρίνει ο καθένα αν τα ιδεολογικά ζητήματα είναι πιο σοβαρά από την ε, διεκπαιρέωση του ζητήματος μέσα στη θητεία. Για την εποπτεία της αγοράς ε, υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση στην οποία βλέπω να μην έχει αποδεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφοροποίηση μεταξύ κινδύνου και συμμόρφωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο να διευκρινιστεί αυτό με σαφήνεια ε, και πρέπει να ξέρουμε σε τι θα εξυπηρετεί το RAPEX, σε τι θα χρησιμοποιείται. Το RAPEX θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καταγράφεται το επικίνδυνο προϊόν. Δεν θα πρέπει να καταγράφεται κάθε πρόβλημα συμμόρφωση, γιατί διαφορετικά δεν θα δώσει αποτελέσματα. Επίση, θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι συμπληρωματικό προς το RAPEX και το οποίο θα περνάει από τη μη συμμόρφωση για τα, πιο, για τα πολύ επικίνδυνα προϊόντα αυτομάτως στο RAPEX. Αλλά πρέπει να είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τα δύο συστήματα. Δεν μπορεί το RAPEX να ενσωματώσει όλα τα προϊόντα. Δεν μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο θα ενσωματώνει τα πάντα. Για τι κυρώσει. Εγώ αποσύρω την ε, τροπολογία μου προς όφελος της δικής σας, ε, κύριε Χέλβεκ, γιατί βλέπω ότι έχει μια πολύ καλή ε, βάση να προσφέρει και μπορεί να αποτελέσει καλή, καλή βάση συζητήσεω. Ένα άλλο θέμα που κρίνω πολύ σημαντικό και εσείς επίσης το αναφέρατε, αν και δεν είμαι σίγουρη το κατάλαβα όπως θα ήθελα στα γερμανικά, ε, το ζήτημα της ε, εμπορίας του προϊόντος, των μεθόδων εμπορίας των προϊόντων, της διάθεσης στην αγορά και της διαφήμισης. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιες μέθοδοι διάθεσης στην αγορά όπως ε, η διαδικτυακή, το διαδικτυακό εμπόριο ή κάποιες άλλες μέθοδοι να βγαίνουν έξω από το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία και να μην επαληθεύεται η ασφάλεια των προϊόντων. Ε, ασφάλεια προϊόντων λοιπόν, εποπτεία Αγορά, ε, Κυρία Σάλτε Μόζερ, θα ήθελα να απευθυνθώ απευθεία σε εσά, γιατί συνεργαζόμαστε στο θέμα αυτό εντατικά και οι δύο έχουμε αισθανόμαστε ιδιαίτερη δυσφορία για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται το ζήτημα αυτό και πάντοτε διαρωτώμεθα πώ είναι δυνατόν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε επιτέλου να υιοθετήσει αυτέ μα τι ανησυχίε και να δώσει ουσιαστική βελτίωση στι ε, προτάσει ε, στον τομέα αυτών. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει και θα συμφωνήσετε μαζί μου, ελπίζω, να πούμε ότι στο ζήτημα του CE, ε, του, του, της Ευρωπαϊκής σήμανσης του Ευρωπαϊκού Σήματος, δίνουμε λάθος εικόνα και παραπλανούμε τον καταναλωτή και ότι θα πρέπει να βρούμε μια ουσιαστική λύση στην υπόθεση αυτή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι μπορώ να δείξω κατανόηση για τα επιχειρήματα που προβάλλονται σε σχέση με το CE+, το, το νέο ευρωπαϊκό σήμα, ε, αλλά πάλι δεν είμαι βεβαία ότι αυτό επιλύει όλα τα προβλήματα, γιατί ούτως ή άλλω ε, τα μη πιστοποιημένα προϊόντα και επικίνδυνα ακόμη κατέληγαν στις αγορές μας με τους ίδιους όρους που κατέληγαν και τα πιστοποιημένα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να βελτιώσει αυτή την κατάσταση το C++ και να προσφέρει ε, ασφάλεια για τον καταναλωτή του. Αντίον ανησυχώ ότι δεν πρόκειται να το καταφέρει. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε και να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, αναλογιστούν το τι σημαίνει αυτό το σήμα, τι μπορεί να συνεπάγεται και ταυτόχρονα να ε, επιφορτήσουμε τη σχετική ευθύνη εκείνου που έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα της εποπτείας τη αγορά. Γιατί μπορεί βεβαίω να έχουμε σαν πρώτο υπεύθυνο τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα, αλλά εάν έχουμε σύστημα επιστοποίηση από τρίτον, δεν μπορεί αυτό να παλάσεται πάση ευθύνη. Εφόσον δίνει το πιστοποιητικό, θα έχει στον ίδιο βαθμό ευθύνη με τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι επίση ότι θα θέλαμε να, ε, θα μπορούσαμε μάλλον να τονίσουμε το ζήτημα ε, με άλλο τρόπο, να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητεί τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης, η απόδειξη ότι η πιστοποίηση ή η η είναι σωστή, αλλά αυτό μπορεί να προξενεί καθυστερήσει. Και το ζήτημα, όλη η λογική πίσω από το σύστημα CE ήταν η ταχύτητα. Ε, πρέπει όμως η εποπτεία της αγορά να ε, ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Λύσεις πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν η μόνη λύση να είναι να ε, καταργηθεί το, σήμα, το ευρωπαϊκό σήμα θα βρούμε λύσεις πιστεύω. Εκεί που θα συμφωνήσω μέσα είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει γρήγορα η ε, ψηφοφορία. Ε, το made in ή country of origin δεν ξέρω κατά πόσον αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ΣΥ, γιατί αν δούμε την, τους χωρισμούς που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την χώρα προελεύσεως, ε, μπορούμε ωραιότατα, για να δώσω ένα πολύ απλό και κοινό παράδειγμα, να δούμε έναν Κινέζο κατασκευαστή ο οποίος ε, φέρνει τα ε, ανταλλακτικά, τα κομμάτια καλύτερα του ε, προϊόντο του σε ένα ευρωπαϊκό κράτο, κάνει μόνο την συναρμολόγηση στην Ευρώπη και μετατρέπει το κατά βάση κινέζικο προϊόν του σε ευρωπαϊκό με, χώρα, με ονομασία προελεύσεω made in και ούτω καθεξής. αυτό νομίζω ότι δεν λύνει κανένα πρόβλημα λοιπόν και πολύ φοβούμε ότι η υπόθεση αυτή και οι εκθέσεις ε, οι δύο κινδυνεύουν στο Συμβούλιο να, ε, να σταματήσουν την πορεία τους. Γι' αυτό δεδομένου ότι έχουμε και χρονική πίεση και θέλουμε να περάσουν αυτές ε, οι νέες προτάσεις, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν είναι πιο σημαντικά τα αισθήματα στο οποίο έχουμε ο καθένα την ιδεολογία του και τις θέσεις του ή αν θέλουμε περισσότερο να βοηθήσουμε ώστε να παράσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Ορισμοί για τους ορισμούς ασφαλώς και χρειαζόμαστε σαφείς και καλούς, ορισμού, ορισμούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε γι' αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή τους ορισμούς της Επιτροπής. Έχω κάνει κάποιες προτάσεις δικές μου, δεν είναι τέλειες, μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επεξεργαστούμε τα θέματα αυτά, γιατί η Επιτροπή δεν έχει κάνει καλή δουλειά στην υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο Άσλι Φόξ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω την κυρία Σαλντεμόζε και τους λοιπούς και οδησηγητές για την εργαστή συνεργασία που είχαμε στο θέμα. Ε, Δυστυχώ ε, δεν άκουσα τι ε, εισαγωγικέ παρατηρήσει ούτε τι δικέ σου τη κυρία Αλντεμόζη, γιατί ήρθε και πέντε λεπτά νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι εσεί ξεκινήσατε πολύ νωρίτερα, γιατί έχασατε μισή συζήτηση. Είμαι πολύ απογοητευμένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, η ομάδα μου οργάνωσε μια δημόσια ακρόαση με καμιά δεκαριά ενδιαφερόμενου και την ΑΝΕΚ με θέμα το, τη σήμανση σε ε, και την σήμανση της ε, προέλευσης. Σε κανένα από τα δύο θέματα δεν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήταν, θα ήταν επωφελές για τον καταναλωτή. Μπορεί να υπάρχουν άλλα ωφέλη, αλλά για τον καταναλωτή το όφελος είναι μηδενικό. Η αναφορά της προέλευσης ε, δεν είναι ε, πραγματικό ωφέλιμο μέτρο, αλλά προστατευτικό. Αν θέλουμε για λόγους προστατευτισμού να το εισαγάγουμε, ναι, αλλά να το πούμε, για, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν είχαμε Αν λέγαμε ότι ήταν για την χρυλασιμότητα, εντάξει, αλλά το μέτρο είναι αμυγό προστατευτικό για να αφορά τη προέλευση και θα αντιταχθούμε. Σε ό,τι αφορά τη σήμανση CE, είμαι ε, διαλλακτικός ε, και μπορείτε να με πείσετε αν έχετε βάσιμα επιχειρήματα ότι είναι υποφελέ για το καταναλωτή. Αλλά από τη στιγμή που κάποιο είναι ικανό να πλαστογραφήσει ένα σήμα σε Ε, γιατί να μην μπορεί να πλαστογραφήσει και ένα σήμα σε Ε. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε την υποπτία τη αγορά, όχι να δημιουργήσουμε ένα νέο σήμα που θα έχει ελάχιστα πλεονεκτήματα. Επανέρχομαι τώρα σε, σε προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα παιδιά ε, και μιμούνται τρόφιμα. Γνωρίζει η κυρία Σχαλντεμόζε τι απόψει μου για το θέμα αυτό, θα τι επαναλάβω. Με την παρούσα διατύπωση πάντω η νομοθετική πρόταση είναι προβληματική. Θα πρέπει να βρούμε μια καλή λύση ώστε μια επιχείρηση ε, που ε, κάνει παρασκευάζει σαπούνι που μοιάζει με κέικ να μην στερείται την δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Οι προτάσεις για τέτοια προϊόντα που μιμούνται τρόφιμα και είναι ελκυστικά για τα παιδιά είναι περιοριστικές και θα πρέπει να τροποποιηθούν. Τέλος, το θέμα των ποινικών κυρώσεων. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να επαφείται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν είναι δέον να επιβάλλουμε εμεί στα κράτη-μέλη, να υποδεικνύουμε στα κράτη-μέλη τι ποινικέ κυρώσει που θα πρέπει να προβλέπουν. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό και θα πρέπει να επαφείται στα κράτη-μέλη. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα τη εποπτεία τη αγορά, Ό,τι αφορά την αρχή τη πρόληψη, πρόκειται για μια αρχή που κατοχυρώνεται στι συνθήκε. Δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε σε κάθε ε, νομοθετική πρόταση μόνο επειδή ε, αρέσει σε μερικού αυτή η αρχή της πρόληψης. Ήδη ε, η, η, η συνθήκη τη Λισαβόνα περιλαμβάνει σε πολλά σημεία πολλέ και διάφορε αρχέ, όχι μόνο της πρόληψη. Δεν χρειάζεται σε κάθε ε, νέα νομοθεσία να τις αναφέρουμε όλες, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν μερικοί. Σε ό,τι αφορά το RAPEX, το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα, συμφωνώ με την κυρία Ρούλε. Αν θέλουμε να είναι χρήσιμο, τότε να περιορίζεται μόνο σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Τώρα, σε θέματα εργαστηρίων, ευρωπαϊκών εργαστηρίων. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να έχει και το δικό της ε, παρατηρητήριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τέτοια παρατηρητήρια, μπορεί να επαφείται σε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται να έχει το δικό της παρατηρητήριο. Τέλος, για τις κυρώσεις. Οι προτάσεις λένε αντίστοιχε ή ανάλογες με το τζίρο, με το κύκλο εργασιών. Γνωρίζετε ότι διαφωνώ. Θα πρέπει να σχετίζεται με τα κέρδη κυρώσεις και όχι με τον κύκλο εργασιών. Και πάλι ε, τα κράτη-μέλη να κρίνουν ένα σκόπιμο να επιβάλλουν είτε ποινικέ κυρώσει είτε οποιοδήποτε κυρώσει πρόστιμα. Τέλο, ε, θεωρώ ότι το πολύ αυτό σημαντικό θέμα χρήζει περισσότερη ε, και πιο σχολαστική μελέτη και περισσότερων συναντήσεων των σχεδόν εισηγητών και θα πρέπει να εκπονήσουμε τι συμβαστικέ τροπολογίε. Λυπάμαι που ξεκινήσατε νωρίτερα το προγραμματιζόμενο τη συζήτηση και έχασα πολλά χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσει, αλλά αν θέλετε να καταλήξουμε σε καλή συμβαστική λύση θα πρέπει να προβλέψετε πολύ περισσότερε συναντήσει με τους κοιόδης ηγητέ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Αλβίνη, ο επόμενος ομιλητής μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Ε, η έκθεση ε, μιλά για την ασφάλεια των προϊόντων. Ε, μερικοί χαρακτηρίζουν την ομάδα μου ως ευρωσκεπτικιστική. Ε, το Μιλάνο και η είναι στην καρδιά της Ευρώπης ε, και είμαστε φιλοευρωπαίοι, αλλά να, να συνεννοηθούμε τι εννοούμε όταν λέμε Ευρώπη, γιατί ο καθένας ε, την προσδιορίζει με διαφορετικό τρόπο. Και αν αρνείται κανεί ότι οι πληροφορίε για την προέλευση και τον τρόπο παρασκευή ενό προϊόντο δεν είναι απαραίτητη, είναι σαν να αδιαφορούμε για την ασφάλεια του προϊόντος. Εγώ έχω ένα δεκάχρονο παιδί. Θέλω ο πολίτη να έχει όλε τις απαραίτητες πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων, των σαπουνιών, των ε, προϊόντων, των παιχνιδιών, των σεντονιών, οτιδήποτε ε, μπορεί να πιάσει ο γιος μου θέλω να είναι απολύτως ασφαλές. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις περιβαλλοντικές και τις συνδικαλιστικές προδιαγραφές, αλλά αυτές δεν είναι οι ίδιες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε και να το να αρνείται κανείς το γεγονός ότι η ασφάλεια δεν σχετίζεται μόνο με τη σαφή αναφορά της χώρας προέλευσης, είναι σαν να αρνούμαστε ότι είμαστε εδώ στις Βρυξέλλες και συζητούμε για το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να ε, θελοτυφλούμε. Ούτε είναι προστατευτισμός αυτό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν παρόμοια μέτρα. Το ίδιο και η Κίνα, η Ιαπωνία, ο Καναδάς. Και αν το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί να έχουμε εμεί δίκιο και οι υπόλοιποι άδικο. Ίσως το αντίθετο συμβαίνει. Ίσως οι υπόλοιποι έχουν δίκιο. Και θα έπρεπε και εμείς να ε, αντί να προστατεύουμε τα δικαιώματα των άλλων, να προστατεύσουμε πραγματικά τους καταναλωτές μας. Επίσης, δεν εκπροσωπούμε μόνο καταναλωτές, αλλά πολίτες που είναι αγοραστές. Και όταν κάποιος αγοράζει, θα πρέπει να είναι σωστά κατατοπισμένος, να ξέρει τι αγοράζει, όποια και είναι η πολιτική του ιδεολογία. Και η Λίγα του Βορρά κατέθεσε μια τροπολογία πολύ πιο φιλόδοξη. Θεωρούμε ότι και για τους αγοραστές αλλά και για τους εμπόρους και για τους παραγωγούς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν από πού προέρχονται οι πιτζάμες ε, που φορούν τα παιδιά τους. Ακόμη και αν η πιτζάμα κατασκευάζεται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό για όλους να γνωρίζουν την προέλευση του προϊόντος. Και για τους παραγωγούς, και για τους διανομής, και για τους εμπόρους, και για τους καταναλωτές γιατί μερικοί παραγωγοί κάνουν τεράστιες επενδύσεις και τεράστια προσπάθεια στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Γιατί να μην αναγνωρίζετε κάτι τέτοιο. Αν επιμείνετε σε αυτή τη θέση, η δική μας ψήφος θα είναι φιλοευρωπαϊκή. Γιατί από τη στιγμή που κοπτόμαστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και να φέρουμε τους πολίτες κοντά στην Ευρώπη, δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε μέτρα που ενισχύουν την ασφάλεια των προϊόντων. Γιατί κοπτόμαστε και για τα περιβαλλοντικά και τα συνδικαλιστικά θέματα και είδαμε στην Ιταλία στι τελευταίε δημοσκοπήσει χαλαρών και μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών και στην Ευρώπη και στα θεσμικά όργανα. Γιατί λοιπόν ο Ιταλός καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη σε μια Ευρώπη που φαίνεται ότι διαφορεί για την ασφάλεια των προϊόντων μια και αδιαφορεί για την προέλευση των προϊόντων. για να υπερψηφίσουμε θέλουμε πιο λογικές λύσεις ε, για όλους και όχι μόνο για ορισμένους. Καλή τύχη σας εύχομαι και στις συγκεκριτές και στην Ευρώπη, αλλά αν θέλουμε εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να αποδείξουμε ότι την αξίζουμε και όλα. ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Περνούμε στους επόμενους ομιλητές. Στάλλαρ Κοφαιράτη και Γκέμπχαρντ έχουμε ακόμα. στον κατάλογο μιλητών. Κυρία Στέλλα. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει τον λόγο, παρακαλώ να μας το πει. Ευχαριστώ κύριε Πίτερ Κάινιον. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συνήθως η δική μας επιτροπή ε, κατά χράτη του χρόνου της τώρα ε, κάνουμε πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε γι' αυτό. Βεβαίω και θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσει ε, με του κοιόδης. Το είπε και η συγγήτρια ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιο είδο συμφωνία, συμβασμού. Βεβαίω θα υπάρχουν ε, σημεία στα οποία δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά συνεργαζόμαστε όσο γίνεται καλύτερα για να βρούμε αυτού του συμβιβασμού. Λοιπόν, αναφερθώ σε μερικά σημεία. Πρώτον, για το RAPEX τον κίνδυνο, το σοβαρό κίνδυνο. Εγώ συνάντησα κάποιους που ασχολούνται με ζητήματα εποπτείας αγοράς την Δευτέρα και εκείνοι λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις και στο Συμβούλιο. Βλέπω ότι εκπροσωπείται το Συμβούλιο εδώ σήμερα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πει το Συμβούλιο τι συζητήσεις διεξάγει για αυτό το θέμα, γιατί ήταν σαφές για μένα ότι υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις, ότι δεν θα υπάρξει σαφήνεια, ε, αλλά και ότι θα, υπονομεύει, θα υπονομευθεί η γνώση των καταναλωτών και η προστασία των καταναλωτών. Έτσι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των ορισμών. Πρέπει να δούμε τι δεν πάει καλά αυτή τη στιγμή. Γιατί σε κάποια κράτη-μέλη αν ένα προϊόν ε, βλάψει ένα παιδί ε, είναι σοβαρό ή αν σκοτωθεί ένα παιδί, αν πεθάνει ένα παιδί δεν είναι σοβαρό. Εμένα με απασχολούν και τα δύο βεβαίως. Ε, και για αυτά τα προϊόντα που αφορούν τα παιδιά και μιμούνται ε, το φαγητό. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει προϊόντα που βλάπτουν τους ευάλωτους καταναλωτές και έτσι χαίρομαι που αναφέρεται σε αυτή την οδηγία το θέμα των ευάλωτων καταναλωτών. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το, για το σήμα, το εμπορικό σήμα είναι θετικό, όμως δεν θα πρέπει να το συζητήσουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Είναι κάτι που θα πρέπει να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Και θέλω να υπάρξει και δράση σε αυτό το θέμα. Thank you. Uh, then... Ευχαριστώ. Κοφεράτη. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστώ και τις δύο συγγήτρες για την πολύ καλή δουλειά που παρουσιάσατε εδώ συνοπτικά, έχουμε να κάνουμε με μία σειρά από προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε στο μέλλον, χάρη στη δική σας συμβολή. Σας έχω κάθε εμπιστοσύνη. Ο δρόμος που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα είναι μακρύς, έχουμε σημειώσει σημαντικές προόδους. Έχω μαζί με συναδέλφους καταθέσει τροπολογίες, για τις οποίες όμως δεν θα κάνω λόγο τώρα. Ήθελα μόνο να φερθώ σε κάποιο σημείο που θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Ο στόχος μας και ο ρόλος και της Επιτροπής μας τελικά είναι να δώσουμε εγγυήσει για τον αγοραστή, για τον καταναλωτή. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι λοιπόν, η αδίποτε πληροφορία μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή και τον αγοραστή θα τους επιτρέψει να επιλέξουν ένα προϊόν με τα λόγου γνώσεως. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ισχυριστεί ότι όσο λιγότερα ξέρει ο καταναλωτής, τόσο λιγότερο κινδυνεύει η υγεία του. Έτσι λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο καταναλωτής να χρησιμοποιεί προϊόντα χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση και κατά τρόπο ανεύθυνο εντό εισαγωγικών, ακριβώ γιατί δεν είναι ενήμερο για κινδύνου που ενδεχομένω ενέχουν τα προϊόντα αυτά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ενημερώσουμε τους καταναλωτές και στον μέγιστο δυνατό βαθμό και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων που μιλούν για ενδείξεις καταγωγής ή προελεύσεως. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει και για τις πρώτες ύλε να υπάρχει αναφορά της προελεύσεως και για τα συστατικά του προϊόντος. Οτιδήποτε δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε καλύτερα για ένα προϊόν. Πρόκειται για ε, πληροφορίες σοβαρές, ουσιαστικές που θα μας επιτρέψουν να ε, επιτύχουμε το στόχο μας που είναι η καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και του ε, αγοραστή. Τι σημαίνει προστατευτισμός εάν βάλουμε ονομασίες προελεύσεως, ο προστατευτισμός στην αδιαφάνεια, στην απουσία διαφάνειας, στην, στις άγριες συνθήκες αγοράς και τον άκρατο ανταγωνισμό επικρατεί. Όταν δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει από πού προέρχεται ένα προϊόν, μπορούμε να μιλούμε για θεμητό ανταγωνισμό. Το αντίθετο ισχύει. Όταν δεν γνωρίζουμε από πού έρχεται ένα προϊόν, αντιμετωπίζουμε τους μεγαλύτερους κινδύνους, που μπορεί να φτάνουν μέχρι και το, το ποινικό δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι σημαντικές οι παρατήσεις, οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν, αλλά θέλω να λαμβάνετε υπόψη η χώρα προελεύσεως ακόμη και για τις πρώτες ύλε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, υπογραμμίζω όχι για λόγους ιδεολογίας, αλλά για λόγους πρακτικούς. Όταν αγοράζω ένα προϊόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρω τι αγοράζω, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω εάν το προϊόν αυτό έχει παρασκευαστεί με τους κανόνες του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ε, κανόνων ανταγωνισμού, των εργασιακών σχέσεων και ούτω καθεξής. Διαφορετικά επικρατεί η αδιαφάνεια και όταν έχουμε συνθήκες αδιαφάνειες μπορεί να συμβεί το κάθε τι. Και βέβαια αυτή την ευθύνη εγώ δεν θέλω να την, να την ε, επομιστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Σε ένα-δύο σημεία μόνο τη συζήτηση, θα επιμείνω και θα αντιδράσω. Είναι ορισμένα από αυτά πολύ σημαντικά. Είμαστε αγορά, είμαστε σήμερα με Επιτροπή της Ιστορικής Αγοράς μένα, αλλά και προστασία του καταναλωτή δε. Και οφείλουμε να μεριμνούμε στο να προσφέρουμε στους καταναλωτές μία αγορά για την οποία μπορούν να αισθάνονται εμπιστοσύνη. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε λοιπόν αυτό. Δύο θέματα που έχουν συζητηθεί πολύ εδώ, το σήμα C καταρχάς και η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως αφετέρου, είναι πολύ σημαντικά σημεία της συζήτησης. Το σήμα CE καταρχάς. Τι είναι τελικά. Δεν είναι σήμα ασφάλειας. Είναι ένα σήμα ε, με το οποίο η επιχείρηση δηλώνει η ίδια ότι έχει τηρήσει τους κανόνες παρασκευής που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποτελεί σήμα ποιότητα στο σήμα ΙΣΥ. Πολλοί όμως είναι οι τη Ευρωπαϊκή Ένωσης λόγω της παραπληροφόρησης, λόγω του ότι υπήρξαν κάποιες εκστρατείε και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, όπως είπε εύστοχα η κυρία Ρούλε, ε, θεωρούν ότι το σήμα αυτό αποτελεί εγγύηση ασφάλεια. Είναι όμω λάθος αυτό. Έχουμε συζητήσει λοιπόν στην Επιτροπή μας αρκετές φορές το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε για το σήμα CE και αυτήν τη διάσταση της ασφάλειας. Και το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αν μπορεί κανείς να παραποιήσει το σήμα, γιατί οτιδήποτε μπορεί να αντιγραφεί και να παραποιηθεί, δεν είναι επιχείρημα αυτό, γιατί είναι τελείως μηδενιστικό και εκμηδενίζει οδήποτε προσπάθεια. Ασφαλώς και μπορεί κάποιος να παραποιήσει να αντιγράψει το σήμα. Αλλά εάν προχωρήσουμε σε ένα σήμα CE+, το οποίο θα ισχύει για ιδιαίτερα σοβαρούς και συγκεκριμένους τομείς, θα έχουμε ένα σύστημα όπου δεν θα επιτρέπεται η πιστοποίηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή εισαγωγέα, αλλά από τρίτο φορέα. Και αυτό προτείνει η κυρία Σάλτε Μόζερ, ε, μια πρόταση την οποία θεωρώ εγώ πολύ σωστή. Και έχει δίκιο η κυρία Ρούλε, πιστεύω, όταν λέει ότι θα πρέπει ε, να μεριμνήσουμε σε περίπτωση που πιστοποιείται κάτι το αναλυθές να μεταφέρεται, να μεταβιβάζεται καλύτερα και η ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε μεταξύ μας οι ομάδες να το συστήσουμε και να το ρυθμίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να απορρίπτουμε εκ προημίου την ιδέα αυτή για να, και να λέμε ότι δεν φέρνει κανένα, ε, καμία πρόσθετη αξία. Ε, το δεύτερο θέμα, η ένδειξη καταγωγής ή προέλευσης. Ξέρω ότι πολλοί πολίτες θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχεται ένα προϊόν, πώς κατασκευάστηκε. Πολλές φορές αυτό αποτελεί και κριτήριο αγοράς για τον καταναλωτή. Ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί καταναλωτές οι οποίοι αδιαφορούν απολύτως. Αλλά εμείς ποιον πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτόν ο οποίος είναι ένας όριμος εντός εγωγικών καταναλωτής και θέλει να ξέρει και με βάση τη γνώση της προελεύσεως αποφασίζει να αγοράσει, να μην αγοράσει το προϊόν αυτό ή όχι. Γιατί σε αυτόν, εάν δεν δώσουμε την, ε, την ε, πληροφορία, ουσιαστικά δεν του επιτρέπουμε να κάνει την επιλογή. Ή αλλιώς υπάρχει λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι να σου πω, και εγώ άμα δω ένα, ένα πουκάμισο το οποίο έχει, ε, έχει, το έχουν υφάνει και ράψει σε κάποια άλλη χώρα ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το φέρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να του ράψουν μόνο τα κουμπιά στη Γερμανία ή την Ιταλία. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι κατασκευαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα μεγάλο περιθώριο για ε, έκτροπα, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθεί το σήμασί. Πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση, το πώς μπορούμε διαφορετικά να το οργανώσουμε και να το ενισχύσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και πρέπει σε αυτό να δώσουμε περισσότερη προσοχή πιστεύω χαιρετίζοντα την παρατήρηση της κυρίας Χάλντε Μόζερ ότι είναι διατεθειμένη να κάνει επιπλέον συναντήσεις με τους σκιώδεις συγκητές προκειμένου να εμβαθύνει και να διευκρινίσει τα εκκρεμίστηματα γιατί θα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα κείμενο καλό, στέρεο, με υποστήριξη στο δυνατόν ευρύτερη, ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει μια καλή και ευρεία βάση διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και το οποίο θα μπορεί να κλείσει μέσα στην τρέχουσα θητεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να καθυστερήσει άλλο το θέμα αυτό και να περιμένουν οι πολίτε και οι καταναλωτέ. Σα ευχαριστούμε. Θέλει άλλο κανεί το λόγο. Κύριε Σόμπερ Μάιερθ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την κυρία Γκέμπχαρτ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσοχή του καταναλωτή να υπάρχει μια σαφής και καθαρή αλυσίδα παραγωγής και κατάληξη στην αγορά ενός προϊόντος. Δεν θέλει να γνωρίζει ένα ε, να έχει μια χονδρική εικόνα της κατασκευής της παραγωγής ενός προϊόντος ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει από πού ε, προέρχεται. Το ε, το μπέικον του Τυρόλου επί παραδείγματι που είναι ένα χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής μου δεν είναι δυνατόν να δεχθώ εγώ να φτάνει, να ξεκινάει από το Βέλγιο ή την Ολλανδία και απλώς όταν μπαίνει στην ε, Αυστρία να παίρνει το χαρακτηρισμό μπέικον ε, Τυρόλου. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτής. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε αυτή την ενημέρωση και τη διαφάνεια στον καταναλωτή. Δεν ε, βλέπω άλλους ομιλητές. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη στην κυρία Δέσποινα Σπανού για να σχολιάσει και κυρίως την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναφοράς και την Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για Τραυματισμούς και το κατά πόσο θα ήταν εφαρμοστεί αυτά τα μέτρα και χρήσιμα. Θέλουμε λοιπόν τις απαντήσεις και στα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση θέλετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω και την κυρία Ελιάνα Μπρίγκμαν δίπλα μου, την Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, θα καλύψει τις σχετικές ερωτήσεις. Έχουμε απαρτία στο επιτελείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα χρήσιμα σας σχόλια. Σημειώνουμε πρώτο με γοργό ρυθμό στο θέμα αυτό. Ήρθα κάπως καθυστερημένα γιατί ήμουν στη συζήτηση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων για το θέμα της, του σήματος προέλευσης, της ένδειξης προέλευσης. Υπάρχει πραγματικά ε, μεγάλη προθυμία και επιθυμία να διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό αυτά τα θέματα και ελπίζω να σας βοηθήσω με κάποια τεχνικά σχόλια να διαλευκάνετε κάποια σημεία και να σημειωθεί πρόοδος και τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα κάποια σχόλια για τα όσα ακούσαμε σήμερα. Ε, ευχαριστώ καταρχήν για τις τροπολογίες. Πρωτορχικός μας στόχος είναι για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα της αγοράς να υπόκειται στις προδιαγραφές ασφάλειας. Γι' αυτό και η πρόταση ε, είναι ένα δίκτυο ασφαλείας. Αυτό θέλαμε. Αυτό είναι ο στόχος που επιτυχάνουμε, εξασφαλίζοντας την ε, εφαρμογή όλων των ε, γενικών διατάξεων ασφάλειας για όλα τα προϊόντα, εναρμονισμένα και μη, και ταυτόχρονα είπαμε ότι δεν θα γεμίζουμε κάποια κενά. Όταν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία, δεν θα πρέπει να έχουμε μια κατάσταση όπου οι οικονομικοί φορείς προσκρούν σε επικάλυψη ή σε πολλαπλασιασμό του γραφειοκρατικού ή διοικητικού άχθους. Αυτά σε ό,τι αφορά το δίκτυο ασφαλείας, σε ό,τι αφορά ε, το σήμα προέλευσης. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το ακούσαμε από πολλούς. Δεν πρόκειται για μια καινούρια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες παγκόσμιας οργάνωσης να έχουν τέτοια νομοθεσία για, το, για την αναφορά προέλευσης. Ε, εμείς δεν έχουμε, αλλά δεν ανακαλύπτουμε το τροχό εδώ είναι ένα σημείο, το σήμα προέλευσης, που το εφαρμόζουν πολλοί άλλοι εμπορικοί μας εταίροι και ήδη το εφαρμόζουν και πολλοί οικονομικοί φορείς μας. Κάποιος ανέφερε ότι ε, κάποια επικίνδυνα προ, προ, προϊόντα μπορεί να μην έχουν αυτή την, ε, το σήμα προέλευσης. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν ανέκαθεν ο καλύτερος εντοπισμός, ε, ταυτοποίηση και χνηλεσιμότητα χάρη ασφάλειας. Γύρω στο 10% των επικίνδυνων προϊόντων που δεν αναφέρονται στο RAPEX είναι προϊόντα που οι αρχές εποπτείας δεν είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσουν την προέλευση αυτών των προϊόντων. Οπότε χωρίς τέτοια στοιχεία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν βελτιώσουμε έστω και κατά 10% την ασφάλεια των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην το κάνουμε και από πρακτική άποψη. Και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε το κόστος. Δεν θεωρούμε ότι είναι αποτρεπτικό το κόστος, ούτε δυσανάλογο ως προς το στόχο της πρότασής μας. Αυτά ως προς το σήμα προέλευσης, την αναφορά προέλευσης. Επίσης, αν μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες τεχνικές πληροφορίες ή βοήθεια, πολύ ευχαρίστως. Σε ό,τι αφορά την αρχή της πρόληψης, που επίσης αναφέρθηκε σήμερα, ε, επαναλάβαμε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συζήτηση την πρότασή μας και την ε, θέση μας ότι η αρχή της ε, πρόληψης είναι ε, βασική αρχή νομικά κατοχυρωμένη και εφαρμόζεται και σε αυτή και σε άλλες προτάσεις. Ταυτόχρονα πολλές χώρες εξέφρασαν την επιθυμία για την μνήμα αυτή τη αρχή. Εναπόκειται στου νομοθέτε να αποφασίσουν αν θα αναφέρεται και στη συγκεκριμένη πρόταση ρητά. Το γεγονό ότι δεν αναφέρεται δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται πάντω, γιατί είναι νομικά κατοχυρωμένη η αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά το σήμα σε Ε+. Διαπιστώσαμε τη διάσταση απόψεων που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και σεβόμαστε την ανάγκη σα να εμβαθύνετε στη σχετική συζήτηση. Πάντω θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο αυτό το σήμα σε Ε+. θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή το κατά πόσο θα επιτρέψει το νέο αυτό σήμα στους καταναλωτές να αντιληφθούν ότι διαφέρει το νέο σήμα C Plus από το προηγούμενο, το CE. Επίσης, δεν είναι κάτι που το έχουμε δοκιμάσει ούτε ελέγξει, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί ε, ένα ενδεχόμενο τέτοιο νέο σήμα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, γιατί από ό,τι ξέρω θα συνεχίσετε τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Τέλος, πολύ σημαντικό όμως θέμα, αναφερθήκατε επανειλημμένα στις διατάξεις για την ειχνηλεσιμότητα και στο RAPEX. Σε ό,τι αφορά το RAPEX, το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα, το κατά πόσο θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε σοβαρούς κινδύνους όπως πρότεινε Αμερική. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντική παλιδρόμη σε σχέση με το στάτο κβο γιατί έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΡΑΠΕΞ. Και μάλιστα όχι μόνο στα θεσμικά όργανα, παντού. Το σύστημα ΡΑΠΕΞ λειτουργεί θαυμάσια. Και πραγματικά δεν βλέπω το λόγο, ούτε μπορεί να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα θέλετε να περιορίσετε το πεδίο εφαρμογή τη. Ε, είπε, είπαν μερικοί ότι δεν θα είναι λειτουργικό. Λάθο Ε, λειτουργεί πολύ καλά, εύρυθμα και θα πρέπει να το βελτιώσουμε, όχι να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή του. Ελπίζω να αλλάξει τη θέση σας προς αυτό. Σε ό,τι αφορά τη βάση δεδομένων για τους τραυματισμούς, αναφέρθηκε από κάποιους ε, ευρωβουλευτέ και αυτό το θέμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες των κρατών μελών να συμβάλλουν σε μια τέτοια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους τραυματισμούς. Θα πρέπει να ελέγξουμε την προθυμία και την ετοιμότητα αλλά και τη βιωσιμότητα το, το κατά πόσο είναι εφικτή μια τέτοια βάση. Δεν διαφωνούμε επί της αρχής, είναι αξιέπαινη η πρόταση αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι και εφικτή και εφαρμόσιμη στην πράξη. Ο λόγος τώρα στη συνάδελφο για τα υπόλοιπα σημεία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες που αφορούν ε, τον κανονισμό εποπτείας αγοράς. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό έργο, το δικό σας και των συναδέλφων σας, για αυτόν τον φάκελο που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Επιτροπή. Εμεί συμμεριζόμαστε αρκετέ απόψει για τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Ε, για παράδειγμα, πολλά ενδιαφέρμενα μέρη και αρχέ υποπτήρες αγορά έχουν αναφέρει ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρξει σαφή ε, διαχωρισμό και διαφοροποίηση μεταξύ των προϊόντων που δεν συμμορφούνται με την ε, εναρμονισμένη νομοθεσία και αφετέρου τα μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα. Για κάποιες τροπολογίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης, ε, με τα χαράς βλέπουμε ότι πολλές ατροπολογίες ε, στηρίζουν ε, οι κανόνες εποπτείας να ισχύουν για όλες τις πωλήσει και τις πωλήσει του διαδικτύου. Επιπλέον, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις που τηρούνται και ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν αποτρεπτικά και επαρκώς και, για παράδειγμα, η πρόταση να συνδεθούν με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ποσό των προσόδων που απορρέουν από την δραστηριότητα αυτή είναι μια ε, καλή πρόταση και θα μπορούσαμε να την εξετάσουμε. Από την άλλη, τουλάχιστον 10%, μια κύρωση του τουλάχιστον 10% επί του κύκλου εργασιών μπορεί να μην επιτρέψει στις ε, αρχές εποπτείας αγοράς ε, να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να διακρίνουν μεταξύ παραβάσεων διαφόρων βαθμών σοβαρότητας και θα ήταν δυσανάλογα υψηλές κυρώσεις ε, για τις μικρότερες παραβάσεις ίσων νοσομασίας. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πολύ ε, από τις προτάσεις της ηγήτριας είναι η αύξηση του συντονισμού ε, σε ό,τι αφορά την εποπτεία των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή είναι εκτεθειμένη να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ κρατών μελών και των αρχών τους για την ε, για τι εθνικέ αρχέ εποπτεία των αγορών και την επίλυση διαφόρων ε, ζητημάτων που ενδεχομένω να ανακύψουν. Υπενθυμίζουμε και τη σημασία στην πρόταση της εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Εποπτεία των Αγορών. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στη συζήτηση για το ρόλο του RAPEX. Δεν θα επανέλθω. Ήθελα μόνο να τονίσω και πάλι ότι ένα σύστημα, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και ότι αυτό το ένα σύστημα θα πρέπει να είναι το RAPEX. Αν κάποια κράτη-μέλη διαμαρτύρονται ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές κοινοποιήσεις, τότε να εξετάσουμε τη συνέχιση, το follow-up που θα πρέπει να δοθεί σε αυτές τις κοινοποιήσεις από τις αρχές εποπτείας επιβεβαιώνουμε ότι το ISC SMS θα είναι ε, θεμελιώδες εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών για έρευνες που διεξάγονται από τις επιμέρους αρχές. Σίγουρα θα συμβάλλει στην ανταλλαγή ε, κοινών πρακτικών και ε, στην αποφυγή των επικαλύψεων που βεβαίω είναι κοστοβόρε. Να καλύψω μερικέ ακόμα πτυχέ. Αφενό έχουμε την πρόταση διαφόρων μελών της Επιτροπής για την εγκαθίδρυση επιπλέον ε, βάσης δεδομένων πανευρωπαϊκής. Κατά τη γνώμη μας, η συμπερίληψη ενός μιας τέτοιας διάταξης στον κανονισμό σε αυτό το στάδιο, χωρίς ε, κατάλληλη τεκμηριωμένη ανάλυση των ε, ωφελών, είναι προώρη και πάλι για την αρχή της αναλογικότητας επιβεβαιώνουμε ότι η πρόταση για την, αγορά, για την εποπτεία των αγορών δεν αναφέρεται στην αρχή αυτή εν γέννη, αλλά προσπαθεί να τη θέσει σε εφαρμογή μέσω επιχειρησιακών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και αρχές εποπτείας αγοράς. Όπως ανέφερε και ένα μέλος της Επιτροπής, είναι κέρια σημασία για όλους τους φορείς στην αλυσίδα εποπτείας αγοράς Χρειαζόμαστε ασφάλεια, βεβαιότητα για το τι θα πρέπει, πρέπει να κάνουν και τι μπορούν να περιμένουν, να προσδοκούν. Κλείνοντας να πω μερικά λόγια για, για το πόσο σημαντικό είναι για την Επιτροπή μαζί με τη δική σας βοήθεια να καταφέρουμε σε συμφωνία με πρώτη ανάγνωση πριν από το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και τι συστάσει του Συμβουλίου, των εκπρόσωπων του Συμβουλίου και θέλω να ρωτήσω τι σχόλια έχει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα για τις δύο εκθέσεις, για τις δύο προτάσεις της Επιτροπής. Αντίστοιχα και στο Συμβούλιο γίνεται πολύ ωραία συζήτηση για τα θέματα αυτά. Οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι. Να ξεκινήσουμε το διάλογο με το Κοινοβούλιο μέσα στη θητεία. Να έχουμε ένα, ένα πρόσκοπτο διάλογο με το Κοινοβούλιο. Σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση. Στο Κορεπές σήμερα έγινε η πρώτη συζήτηση για την προστασία των καταναλωτών. Άρχισε λοιπόν στο επίπεδο αυτό. Και προσωρινά θα μπορούσα να δώσω μια, ερω... μια απάντηση σε μια ερώτηση που νομίζω απευθυνόταν στο Συμβουλίο για τη ΡΑΠΕΞ. Μπορώ να πω το εξής, ότι όντως είναι προσυζήτηση το να μείνει το ΡΑΠΕΞ, ε, να γίνει το ΡΑΠΕΞ στη βασίδα που αφορά μόνο τα επικίνδυνα προϊόντα, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό και μένουν εκκρεμή. Επομένως, άλλο περισσότερο δεν μπορώ να πω. Παρακολουθούμε την ε, ε, υπόθεση και τη συζητούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Άλλα σχόλια, παρατηρήσεις. άλλος. Ναι, κυρία Στάιλερ, ε, θέλετε να μου πείτε τι είδους χρονοδιάγραμμα έχετε, μια και λέτε ότι το έχετε προσυζήτηση στο θέμα, τι χρονοδιάγραμμα έχετε προβλέψει. Πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση. Πότε θα το προβλέψετε στην ημερήσια διάταξη των εργασιών σας. Να γνωρίσουμε και εμείς τι κάνετε. Ναι, ευχαριστώ. Τον Οκτώβριο αναμένονται κάποιοι γύροι διαπραγματεύσεων. Με στόχο να ξεκινήσει ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στο έτος. Για να κλείσουμε το θέμα μας στη θητεία. η Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις, να ακούσουμε την κυρία Σχάλντα Μόζαρ. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια. Η πολύ καλή συναδέλφος Κάθριν Στάιλερ μου είπε ότι θα πρέπει να περιοριστώ στις δικές μου θέσεις να δώσω τις απαντήσεις ε, μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί κάναμε τον Ιούλιο μια τόσο ευχάριστη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών και νόμιζα ότι είχαμε τεράστιο πεδίο συμβασμού, γιατί φαίνονταν όλοι διατεθειμένοι να πλησιάσουν ένα τον άλλον ε, με πολύ καλή διάθεση κτλ. Με τη συζήτηση που είδα σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είμαι τόσο βέβαιη πια. Και θεωρώ ότι κάποιοι συνάδελφοι ήταν αρκετά σκληροί και έδειξαν λίγη διάθεση για συμβασμού. Μάλιστα κάποιοι απεχώρησαν ήδη και δεν ε, κάθισαν καν να ακούσουν τι έχω να του απαντήσω. Αλλά το προσωπικό του φαντάζομαι είναι εδώ και παρακαλώ να σημειώσει και να μεταφέρει το εξή. Εάν μα δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν από το πέρα τη θητεία, για να το καταφέρουμε θα πρέπει ο κάθε ένας να συμπράξει και ο κάθε ένας να υποχωρήσει σε ορισμένα ζητήματα που μπορεί να θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά ιδεολογικά ο καθένας. Και επίσης θέλω να πω το εξή. και για να είμαι σαφής και περιφράστη, εγώ δεν έχω κανέναν ενδιασμό να φτάσω στις ευρωεκλογέ με θεματολογία την ασφάλεια των προϊόντων και να καταγγείλω ποιος υπερασπίζεται και ποιος δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα του καταναλωτή στην Ευρώπη. Δεν με νοιάζει εμένα η υπόθεση αυτή περισσότερο, γιατί είμαι βεβαία ότι μπορώ να εξηγήσω στον καταναλωτή στην Ευρώπη ποιος πραγματικά προσπίστε τα συμφέροντά του. Πολύ απλό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση πολλά, σε πολλά θέματα. Και πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Αν και σημειώνω ότι θα πρέπει να επιδείξουν όλη την ίδια διάθεση για εξέβρεση λύσεων. Εγώ θα το πράξω από πλευρά μου. Εγώ δεν θα δείξω ε, στάση αμετακίνητη σε κανένα θέμα. Εκτός από τις κόκκινες γραμμές βέβαια που έχω ορίσει και θα ήθελα να επαναλάβω ένα πράγμα τουλάχιστον ότι οθετήσαμε τη δέσμη για τα αγαθά πριν από μερικά χρόνια, όπου μιλήσαμε ξεκάθαρα για το ζήτημα των οικονομικών φορέων και αυτό για μένα αποτελεί κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται να υποβαθμίσω την ευθύνη και τις, ε, ευθύνες, καλύτερα των οικονομικών φορέων. Διότι υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει ξεκάθαρα για το, ποιο, το ποιος έχει ευθύνη όταν παίρνει ένα προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά. Πέραν αυτού, είμαι δετεθειμένη να συζητήσω και να υποχωρήσω προκειμένου να βρεθούν λύσεις και περιμένω να γίνουν και προσοχή συνεδρία με του δυσκιώδες συγκεκριτέ, για να βρούμε λύσεις καλές. Και η αγορά μας και οι καταναλωτές μας αξίζουν μια καλή λύση, μια καλή δέσμη μέτρων για την προστασία της αγοράς, για να έχουμε μια καλά λειτουργούσα και ασφαλή εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Πιατικάινεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τους και ηγητές, την συνεισηγήτρια, τη συνάδελφη συγγήτρια καλύτερα, για το, τη δουλειά σε όλη αυτή την υπόθεση. Περιμένω και εγώ να γίνει ο προσεχής γύρος διαπραγματεύσεων και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές λύσεις και υψηλή προστασία για τους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν κλείνουμε τα θέματα 13 και 14 της ημερησίας διατάξεως και το μικρόφωνο της ομιλήτριας. It stands at the moment the consideration of... Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες. 14 Οκτωβρίου Επιτροπή Εσωτερική αγορά 17 Οκτωβρίου για την έγκριση. Θα κάνουμε σκληρή δουλειά γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Και παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι κάποιοι θα χρειαστεί να αποχωρήσουν, αλλά παρακαλώ να μείνετε όσο δυνατόν, να φύγετε όσο δυνατόν πιο ήσυχα για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στο σημείο 15, την Ευρωπαϊκή τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Έχουμε τσέρφο γκάλμπελς εδώ. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε δύο λεπτά. Sorry to disturb you, but uh, could you move up with the discussion? Σας παρακαλώ τις συζητήσεις σας ε, στο διάδρομο. Προσπαθούμε να κλείσουμε κάποια θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Ιλντικό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ευχαριστώ Ξαναμιλάω για τη γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση. Στην άμυνα θα είμαι πολύ σύντομη. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο απευθύνουμε στην, στην Υποεπιτροπή Άμυνας αρμόδια για θέματα άμυνα, η οποία συνεργάζεται με την Επιτροπή Βιομηχανία. Η Επιτροπή Ιστορική Αγορά είναι η δεύτερη που αναλαμβάνει γνωμοδότηση και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι κύριος στόχος της ευρωπαϊκής, της βιομηχανικής ε, και τεχνολογικής βάσης ευρωπαϊκής άμυνας είναι βέβαια να εξασφαλίσει τη, τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και την ασφαλεία τους. 33 είναι τροπολογία συνολικά. Τις καλωσορίζω. Νομίζω ότι προσθέτουν αρκετά προσθέτουν αρκετά στο κείμενο. Θα προσπαθήσω να τι αναδιοργανώσω. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να σημειώσω ότι προηγούμενες προσπάθειες για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αναθεώρησης ευρωπαϊκής άμυνας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού της Ευρωπαϊκής Αγοράς Άμυνας και να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα σχεδιασμού. Ε, βέβαια αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την παρούσα γνωμοδότηση. Μεν μπορούμε ωστόσο να αναλάβουμε βήματα προς την κατεύθυνση, ιδιαίτερα αν επικεντρωθούμε στις δημόσιες προμήθειες. Στην Επιτροπή μας Έχουμε αρκετή εμπειρία και ως εκ τούτου κατατέθηκαν και αρκετές τροπολογίες για τις οποίες θα αναζητήσουμε συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 81 του 2009 προκειμένου να τηρήσουν τις προδιαγραφές για τις δημόσιες προμήθειες στον χώρο της άμυνας. Και παρακαλώ την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση ισότιμων συνθήκων πρόσβαση στην αγορά άμυνας και να περιορίσει τις δυσανάλογες πράκτικες που επικρατούν ορισμένες φορές. Σημαντικό επίσης είναι να μιλήσουμε για νέους τύπους ε, προμηθειών Δέχομαι και υποστήριζω την σχετική τροπολογία του κύριου Χάρμπορ. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τη χρήση των νέων μεθόδων προμηθείων και στην άμυνα και αναφέρομαι εδώ στην, ε, στην ε, προμήθεια πριν από τη διαθέση στην αγορά, εξέταση συγκεκριμένων όρων, χρήση της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής, θέσπιση κινήτρων, μείωση του διοικητικού φόρτου. Και θα επιμείνω στην προμήθεια πριν από την εμπορευματοποίηση ενό προϊόντος γιατί είναι πολύ σημαντική πιστεύω αυτή για τη γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό για να διευκρινίσουμε τα ζητήματα. Και περνάω στην ε, συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Ασφάλειας και Άμυνας και της Επιτροπής μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη θέσή μας για να ε, καλύψουμε και μικρότερα κράτη, αλλά και για να αντιστρέψουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Το Συμβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει στην ε, ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου τα θέματα αυτά προς συζήτηση και πάνω απ' όλα θα πρέπει να δοθούν κατάλληλοι πόροι και για την ε, έρευνα και για την προαγωγή εταιρικών και συνεταιρικών σχέσεων. Έχουμε κάποιες τροπολογίες για την τυποποίηση. Η διαμόρφωση ομοιόμορφων μέσων για την άμυνα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ομοιόμορφης αγοράς άμυνας, αλλά και για την εξασφάλιση λειτουργικότητας. Είναι φυσικά πολύ σημαντικό να συλλέγονται και να αναπτύσσονται από κοινού έργα με διαλειτουργικότητα. Είναι κατά τη γνώμη μου οι συνθήκες αυτές ε, που έχουμε τώρα και οι προδιαγραφές που έχουμε ικανοποιητικές δεν χρειάζεται να εισαχθούν νέε προδιαγραφές. Το θέμα βεβαίως είναι από τα πιο λεπτά, αλλά θα υπογραμμίσω ότι δεν είναι τόσο εκτός των αρμοδιότητων της Επιτροπής μας. Κάθε δε νέα προδιαγραφή μπορεί να περιπλέκει την αγορά Τη Άμυνα. Γι' αυτό έχω κάνει τροπολογία σχετική με, την, ε, με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και βεβαίως μας έθεσε σε κάθε συζήτηση. Εν τέλει, θα ήθελα να αναφέρω την πρακτική ορισμένων κρατών μελών που δίνουν προτεραιότητα στην ε, χώρια ε, βιομηχανία όπλων αμυντική βιομηχανία και προκειμένου να διασφαλίσουν ε, θέσεις εργασίας για τον, τον ε, οικείο πληθυσμό, αλλά και για να διαφυλάξουν το απόρριτο. Και έτσι δεν υπάρχει πρόσβαση για τα λοιπά κράτη, ε, για, για τους κατασκευαστές των λοιπών κρατών, στην αγορά άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ε, υπάρχουν εμπόδια δε που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και ελπίζω η αγορά, η, η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή να βοηθήσει στην αποδιάρθρωση των περί των προσκομμάτων. Έχω προετοιμάσει ήδη κάποιες προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες. Σε μια πρώτη μορφή μόνο. Τις έχετε λάβει πιστεύω. Αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτές. Μπορούμε με τη συζήτηση να τις ε, ολοκληρώσουμε φυσικά με στη θέση των συναδέλφων για περαιτέρω συζήτηση. Είμαι ε, έτοιμη να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και για δίποτε αιτήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Από Σκιώδης έχουμε την κυρία Γκέπχαρτ και τον κύριο Μπιέλαν. Κανονικά περιμένουμε και τον κύριο Σαλβίνη. Έχουμε και τον κύριο Σμιτ. Uh, uh, uh, θα ξεκινήσουμε με την Εύελεν Γκέφχαρτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Πολύ καλή η βάση που μας προσφέρει και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη διάθεση που δείχνει για επεξεργασία συμβαστικών τροπολογιών. Πρόκειται για ένα θέμα όχι τόσο εύκολο, το ξέρουμε. Ένα θέμα το οποίο, ε, στο οποίο αντιδράμε ιδιαίτερη ευαισθησία και ο πολίτης της Ευρώπης. Ελπίζω να μπορέσουν να γίνουν ε, δεκτές ε, οι τροπολογίες μας από όλους συναδέλφους, ειδικά εκεί όπου αναφερόμαστε στη διαφάνεια στις αναθέσεις για παραγωγή προϊόντων από την αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα εκεί όπου η συνεργασία, η σύμπραξη σε ένα έργο μπορεί να μειώσει τις δαπάνες, τις κρατικές δαπάνες στον τομέα αυτών και να οικονομήσει, να εξοικονομήσει πόρους για το δημόσιο κορβανά. Σε αυτό δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα, ειδικά βέβαια ε, είδαμε στη Γερμανία πόσο γρήγορα κατασπαταλήθηκαν χρήματα με την υπόθεση των ε, ε, drones, των ε, μη επανδρομένων αεροπλάνων και πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία. Οι τροπολογίες, οι συμβαστικές 1, 2, 3 που έχω δει μας ικανοποιούν, τις υποστηρίζουμε όπως έχουν. Για την συμβαστική τροπολογία 2 έχω μια ερώτηση, μάλλον 3 λέει ο μιλήτρια, για την ε, προσυμβατική ανάθεση. Πώς το βλέπετε αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ότι η ομάδα μου έχει πολύ επικριτική στάση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με διαφάνεια. Εάν έχουμε δηλαδή μία ε, συζήτηση και προσδιορισμό συνθήκων για μια ανάθεση πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, προφανώς έχουμε πρόβλημα διαφάνειας, αυτό δεν θέλει να συμπράξει η ομάδα μου, το κύριο μας μέλημα είναι η διαφάνεια. Εκεί που ενδέχεται να μην σας ακολουθήσουμε είναι κάποιες τοποθετήσεις και τροπολογίες που ενδεχομένω να τείνουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό διαφωνούμε. Γιατί στόχος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλωστε είναι καταγεγραμμένος και στην Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο ακριβώς τιμηθήκαμε με το βραβείο Ειρήνης, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, είναι ακριβώς να μην επενδύουμε στον πόλεμο, στην τεχνολογία της άμυνας, στην πιο υψηλή τεχνολογία. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή θα είναι η θέση της πολιτικής μου ομάδας. Diesen Änderungsanträgen, auch nicht äh, ähm, Είμαστε πάντως ε, διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε τις συμβαστικές αστροπολογίες εκεί όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη προσθεμένη αξία, περισσότερη ουσιαστική υποστήριξη στην ε, παρασκευή προϊόντων ε, στον χώρο αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Σμιτ για τους φιλελευθέρους ε, κανονικά προηγήσε. Δεν σε είδα πριν στο κατάλογο, συγγνώμη. Ε, είμαι μικρούλης. Μικρός όμως. Δεν φτάσεις εσύ. Όταν και ο Νόμπελ φαίνεται ε, ε, τη δυναμίτιδα άρχισε να τύπτεται από, από ε, ε, άρχισε να τον τύπτει η συνείδησή του και για να εξηλωθεί κάπως θεσμοθέτησε τα βραβεία Νόμπελ. Θέλουμε μια πιο ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία. Κανένα πρόβλημα. Μάλιστα η ομάδα μου κατά πάσα πιθανότητα θα εγκρίνει και τις τρεις σας συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα και θέτω παρεμπιπτόντως και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την εισαγωγή αυτού του μέτρου, ενώ στην Ευρώπη έχουμε παντού μέτρα λιτότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι τι θέλουν οι πολίτες. Θέλουν περισσότερες δαπάνες για τις συντάξεις τους, όχι για την ε, αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Ναι, βέβαια, το θέμα είναι ευρωπαϊκό και αναφέρεται και στη συνθήκη και κατά πάσα πιθανότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες αφιβολίες. Αυτές όμως είναι οι προσωπικές μου επιφυλάξεις. Γιατί θεωρώ ότι αν συγκρίνουμε τις ευρωπαϊκές δαπάνες με τις αμυντικές δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών ή αν συγκρίνουμε με τις αμυντικές δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού, τότε έχω πρόβλημα με την πρώτη σας συμβαστική τροπολογία που λέει ότι θέλουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Εν πάση περιπτώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι συνάδελφοι από την άλλη δεν θα σας υποστηρίξουν. Τώρα για τις υπόλοιπες τροπολογίες δεν έχω πρόβλημα κατέθεσε και μια τροπολογία για την απελευθέρωση των προμηθειών και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις για τα πιο ευαίσθητα προγράμματα και ο κατακαιρματισμός βλάπτει την ευρωπαϊκή αγορά και εθνικές προστατευτικές πολιτικές βιομηχανικές ε, φαίνεται ότι επιτρέπονται από το άρθρο 346 της συνθήκης. Αυτό όμως είναι παρερμηνία του σχετικού άρθρου που ήταν τόσο ευρέω διαδεδομένη ώστε και μετά από μη ευαίσθητες δημόσιες βάσεις ε, στο, ε, υιοθετήθηκε. Για παράδειγμα, υπηρεσίε καθαρισμού, παροχή τροφίμων αποκλείστηκαν από του κανόνε δημοσίων προμηθειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσίων συμβάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είχαμε και προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της παρερμηνίας αυτής. Γι' αυτό και κατέθεσε και τροπολογία. Γενικώ πάντως, δεν έχουμε πρόβλημα με τη γνωμοδότησή σας, κυρία Πέλτς. Θα την υποστηρίξουμε και όταν ήμουν μικρός και υπηρετούσα στην κυβέρνηση της Σουηδίας, ε, είχαμε ε, αρκετά μεγάλο αμυντικό κλάδο που προσπάθησε να μας, προσπαθούσε να μας προστατεύσει από τους γείτονες, όχι βέβαια τη Φιλανδία. Ε, χάσαμε τη Φιλανδία το 1809. Πάντως, τα αντισταθμιστικά ωφέλη που αναφέρατε. Προσπαθήσαμε να πουλήσουμε όπλα στην Ουγγαρία με αντισταθμιστικό όφελο να αγοράσουμε ντομάτε από τη χώρα αυτή. Δεν είμαι 100% σίγουρο, αλλά αυτό θυμάμαι. Αν μπορέσουμε να καταργήσουμε τα αντισταθμιστικά ωφέλη, θα ήταν ε, ευχής έργο για μια πιο αξιοπρεπή αγορά στον αμυντικό κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε τώρα με το ECR. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιέλαν εκπροσωπώ εδώ τον Μάλκομ Χάρμπορ, που είναι ο σκιώδης συγητής. Ο Μάλκομ κατέθεσε δύο τροπολογίες στη γνωμοδότηση της κυρίας Πέλτς. Η πρώτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορά τη τη διαδικασία της νέας ε, εταιρικής σχέσης καινοτομίας ε, στην αναθεωρημένη οδηγία για τι δημόσιες ε, συμβάσεις να τη μεταφέρουμε και στην οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα τη άμυνας όταν αναθεωρηθεί το 2016. Πρόκειται για την τροπολογία 15 του κυρίου Χάρμπορ. Συμφωνώ ότι με την νέα αυτή διαδικασία θα βοηθήσουμε την αμυντική βιομηχανία κυρίως ε, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τις προωθούν. Ελπίζω και χαίρομαι που τελικά συμφώνησε με την τροπολογία αυτή του κ. Χάρμπορ, η συγκεκριά. Η δεύτερη τροπολογία του κ. Χάρμπορ είναι η 13 για τις καινοτόμες ε, πολιτικές, τεχνικές δημοσίων συμβάσεων, προσυμβατικές δαπάνες και ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις για ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ακούσαμε τι επιφυλάξει των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Προ το παρόν δεν έχουμε καταλήξει συμβαστική λύση προκειμένου να παραμείνει η μνήμα στι πρόσυμβατικέ δαπάνε ω καινοτόμο τρόπο δημοσίου συμβάσεων στον τομέα τη Άμυνα. Λυπούμαστε για τη διαφωνία αυτή των σοσιαλιστών, ιδιαίτερα γιατί τέτοιου είδου τεχνικές προσυμβατικών δαπανών είναι πολύ καινοτόμο εργαλείο και αναγνωρίζεται και στο τελικό κείμενο του, της νέας οδηγίες που θα υιοθετήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο. Κατά τη γνώμη μας, προσυμβατικές δαπάνες ε, θα δώσουν όθηση στην τεχνολογική και βιομηχανική βάση της άμυνας ε, και επίσης θα ε, δώσουν ενάψματα και καινοτόμες εταιρικέ σχέσεις. Έχω καταθέσει και εγώ δύο τροπολογίες. Η πρώτη μου αφορά τη χρηματοδότηση σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, στα κράτη-μέλη η σχετική πρόοδος βοηθά σε πολλές βελτιώσεις και σε άλλους καθημερινούς τομείς, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές εφευρέσεις του στρατιωτικού κλάδου στην καθημερινότητα, στο ίντερνετ για παράδειγμα, στο διαδίκτυο. Και επίσης ε, συμφωνούμε για συντονισμένη δράση για να αποσοβήσουμε τις απειλές στον κυβερνοχώρο που ε, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ε, υπηρεσίε ε, του διαδικτύου. Σα ευχαριστώ και ελπίζω να υπερψηφίσουμε την γνωμοδότηση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ του και διηγητέ. Δεν ξέρω αν θέλει άλλο κανεί το λόγο. That is not the case. Uh, yes, uh, Mr. please. Ο κύριο Thank you Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γιατί σε ένα τόσο σημαντικό θέμα η συζήτηση γίνεται ή πρέπει να γίνει με τόσο συνοπτικές διαδικασίες. Εκπλήσω Δεν ψάχνω να βρω το γιατί. Και Βλέπω ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει σωστές προσεγγίσεις. Εντάξει, μπορεί αυτό να το κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Κοινή αμυντική πολιτική στο πρώτο σημείο ίσως δεν είναι τόσο ενδιαφέρον. Απελευθέρωση των δημοσίων προμηθειών και όλα αυτά. Πολύ καλά μέχρι και αλλά αυτό που δεν βλέπω είναι συγκεκριμένες διατυπώσεις. Και όταν είναι τόσο ασαφής διατυπώσεις ή θα καταλήξουμε σε προβλήματα ή θα φτάσουμε σε κάτι το οποίο τελικά μπορεί να μην ήταν καν η πρόθεση της προτάσεως. Όταν, για να δώσω ένα παράδειγμα, ε, προτείνεται να υπάρχει ενημέρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας πέραν των συνόρων κτλ. Πολύ καλά. Αλλά πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε και να εξυπηρετήσουμε τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά που επίση αναφέρεται ότι υπάρχουν και πρέπει να διαφυλαχθούν. Δεν πρέπει αυτό να τα λησμονούμε τα χαρακτηριστικά τη εθνική αμυντική βιομηχανία. Επίσης να γίνεται λόγος για καινοτόμε μεθόδους αναθέσεως και διαγωνισμών. Χωρίς καμιά διευκρίνηση, πάλι μου φαίνεται πολύ ασαφές. Δεν βλέπω πού τίνει, τι επιδιώκει. Είναι πολύ, πολύ ασαφές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν με τόση ταχύτητα. Δεν βλέπω να έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε στην ουσία του τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να στραφώ προς την Επιτροπή. Ο κύριος Ανσιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κατά μέλη της Επιτροπής για τις παρεμβάσεις τους. Από πλευρά τη Επιτροπή είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι πολλέ από τι παρατηρήσει και τι τροπολογίε ανταποκρίνονται ε, στην προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στην ανακοίνωση του Ιουλίου. Ουσιαστικά θέλουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της αγοράς και του βιομηχανικού κλάδου του κλάδου βιομηχανία και τη άμυνα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα εύρωστο ε, νομικό πλαίσιο. Χαιρετίζουμε λοιπόν το γεγονό ότι και πάλι υπογραμμίζεται πώ χρειαζόμαστε μια πραγματική, πραγματικά αποτελεσματική εφαρμογή του κεκτημένου, ιδιαίτερα ό,τι αφορά την οδηγία περί δημόσιων προμηθειών για να αυξηθεί η διαφάνεια των αγορών Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μια ε, βιομηχανική πολιτική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της αν θέλετε. Χρειαζόμαστε τις κατάλληλες δεξιότητες, τα κατάλληλα εργαλεία για να δούμε τι ακριβώς μας χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να τονίσω κάτι που αναφέρεται σε κάποιες τροπολογίες, σε σημασία της τυποποίησης και πιστοποίησης για μας ε, η φυστάμενη έλλειψη κοινού συστήματος πιστοποίησης και τυποποίησης είναι το, ένα μεγάλο εμπόδιο για τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Και αυτό επηρεάζει και την, αποτελεσματικότητα, την ε, ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία. Θα θέλαμε λοιπόν μια καλύτερη προσέγγιση σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα στην πιστοποίηση. Και έτσι θα ε, εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα στην ανάπτυξη νέων ε, προϊόντων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ανάλυση που έγινε, νομίζω ότι εν γέννη συμμεριζόμαστε τόσο υπόθηκαν και εκφράστηκαν και σε τροπολογίες. Ίσως μία παρατήρηση ακόμα που αναφέρθηκε πολύ σωστά. Πράγματι βρισκόμαστε εν καιρό λιτότητας, όμως αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι ότι Ίσως είναι δύσκολο να μιλάμε για αύξηση των δαπανών στις, ε, στην άμυνα. Εμείς όμως τονίζουμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να, ε, να καταστήσουμε τις δαπάνες μας πιο αποδοτικές και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Με των κοινών προμηθειών, μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ ε, πολιτικής προστασίας ε, και στρατού. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θέλω να δείξω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Για το χρονοδιάγραμμα, η ψηφοφορία θα γίνει στις 13 και τώρα για το κλείσουμε να δώσουμε τον λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, για τις παρατηρήσεις σας Είμαι πεπισμένη ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και βεβαίως θα λάβω υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν. Θεωρώ ότι είχαμε τις θα έχουμε τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις εντός του χρονοδιαγράμματος, αλλά ξέρετε ότι είναι πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να χειριστώ τις διαπραγματεύσεις ε, μέσα εντός της προθεσμίας και αν με χρειάζεται βεβαίως είμαι ε, οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Και είμαι σίγουρη ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και εγώ θα ενημερώσω τους κοιόδης σε ό,τι φορά αυτή τη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το τομέα, όμως νομίζω ότι θα πρέπει ε, να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και έτσι να χειριστούμε τις τελικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Καλή τύχη στην εισηγήτρια και στους στους εισηγητές, γιατί δεν έχετε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ για τις επικοδομητικές σας παρατηρήσεις. Κλείνουμε το σημείο 15. Έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής της διάταξης. Κυρίσω λοιπόν το πέρας ε, των εργασιών μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ελπίζω να έρθετε ανανεωμένοι και ξεκούραστοι αύριο. Καλό βράδυ.